Hello everyone. We Αρχίζουμε λοιπόν με το πρώτο θέμα για το απόγευμα που είναι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Η εισηγήτρια είναι η κυρία Γκαρτίνη για αυτό το θέμα συναπόφασης. Σήμερα θα δούμε την, το προσχέδιο εκθέσης όταν είσαστε έτοιμοι, μπορείτε να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι πολύ γεμάτες οι και είχα ένα ε, ραντεβού στο άλλο μέρος, στην αντίθετη πλευρά του κτίριου. Θα προσπαθήσω να σας δώσω μία ανακεφαλαίωση γιατί η πρόταση της Επιτροπής είναι γνωστή. Ξέρουμε την αιτιολογική σκέψη και για αυτή τη φορά δείξαμε στο Κοινοβούλιο ποιοι είναι οι απότεροι στόχοι. Είναι πολύ συνεκτική η έκθεση. Θα ήθελα να σας πω ποιες είναι οι βασικές αλλαγές σε σχέση με την αρχική πρόταση ως προς τη δική μου έκθεση για να ενισχύσουμε το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής, γιατί όλοι θέλουμε έναν πιο εύρωστο μηχανισμό, ο οποίος να δίνει σαφείς ε, λύσεις και ευφύς λύσεις. Ως προς το Rescue, Ξέρετε ότι είχαμε προτείνει έναν απογραφικό κατάλογο. Στην έκθεσή μου έχω αντικαταστήσει τον κατάλογο των μέσων με κατάλογο κινδύνων στους οποίους θα μπορέσουν να ανταποκριθούν τα μέσα για να είμαστε πιο ευέλικτοι και να δούμε και τις τεχνολογικές αλλαγές και εξελίξεις του τομέα όσον αφορά διακόπτει η ομιλήτρια και ξαναπιάνει την πρότασή της από την αρχή. Όσον αφορά ορισμένες προτάσεις του Συμβουλίου, ξέρω ότι ένα από τα κρίσιμα σημεία για το Συμβούλιο είναι η εποπτεία του ρέσκιου και αυτό είναι και το σημείο καμπής αυτής της πρότασης, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις και πόροι. Γιατί αυτή είναι η ανησυχία ορισμένων κρατών μελών. Ας πούμε στην Ιταλία οι πυροσβέστες μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό. Άρα θα βασιστούμε σε επιπρόσθετους πόρους πέρα από αυτούς που προϋπάρχουν και ανήκουν στα κράτη-μέλη. Αυτό ελπίζω να μας βοηθήσει για να επιλύσουμε ζητήματα ορισμένων κρατών Επίσης, πέρυσι το καλοκαίρι χρειάστηκε να βοηθήσουμε χώρες γιατί δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές και τους εμβρισμούς. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να ανταποκριθούμε και να αποστείλουμε δυνάμεις στην Πορτογαλία και όχι στην Ελλάδα ή την Ιταλία και αντιστρόφως. Διαφορετικά μπαίνουμε στην καθαρά κρατική λογική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, επίγουσες ανάγκες. Επίσης, η Επιτροπή δεν αναφέρεται στη χρηματοδότηση του 55% όσον αφορά τις μεταφορές. Και εδώ μιλούμε για πιστώσεις υποχρεώσεων υπό την έννοια ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουν ένα μητρό όπου όλα αυτά τα ε, μέσα να ενταχθούν σε ένα μητρό, γιατί ξέρετε ότι για την πολιτική προστασία θα πρέπει τάχιστα να γνωρίζουμε τι μπορεί να γίνει και τι είναι χρήσιμο. Και η απώλεια χρόνου είναι και απώλεια ζωής. Απώλεια ζωής, απώλεια πολιτιστικής κληρονομιάς και ούτω καθεξής. Θέλουμε λοιπόν επικαιροποίηση αυτού του Μητρώου, όπου φυσικά τα κράτη-μέλη θα ανταποκριθούν με τις διάφορες ε, υποδομές διαχείρισης. Ένα άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την πολιτική προστασία και το Εράσμους είναι ένα Εράσμους για την πολιτική προστασία, έτσι ώστε να συνεισφέρει σε μια ομογενοποίηση της Ευρώπης. Ξέρετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Γιατί θέλουμε να έχουμε κοινέ προδιαγραφές και γι' αυτό θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στη συνέχεια, στο άρθρο 6 της πρότασης υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο, η διαχείριση κινδύνων. Γνωρίζετε ότι κατά την προηγούμενη θητεία είχαμε φτάσει σε ένα συμβιβασμό, ώστε τα κράτη να μην αποτιμούν ε, ολοκληρωμένα τον κίνδυνο, αλλά να το δουν ε, συνθετικά το όλο ζήτημα. Για να λάβουμε υπόψη την ε, διαφορετικότητα και τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη πολλές φορές είναι επιφυλακτικά ως προς την διαβίβαση δεδομένων. Σε αυτή λοιπόν την ε, συγκεφαλαίωση θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα βασικά στοιχεία που διέπουν το κάθε κράτος μέλος, στοιχεία τα οποία όμως να είναι συγκρίσιμα μεταξύ των διαφόρων κρατών. Υπάρχουν και άλλα σημεία όπου ενίσχυσα από την προηγούμενη φοιτεία στοιχεία και σημεία που μας είχαν βρει σύμφωνους σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές, κατά πόσο είναι ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές και επίσης για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, διότι οι πυρκαγιές προκαλούν το 20% παγκοσμίως των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και θα πρέπει να υπάρχει και η περίφημη επικουρικότητα Και εδώ ενισχύουμε και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές μέσα στα πλαίσια της αρχής της επικουρικότητας για την πολιτική προστασία. Αυτά είναι τα βασικότερα σημεία. Υπάρχουν πολλές σημαντικές συνεισφορές γιατί υπάρχουν πολλά κεφάλαια, ας πούμε η διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου. Αυτό θα το δούμε με τους συναδέλφους. Επειδή γνωρίσαμε αυτές τις επίγουσες ανάγκες πέρσι το καλοκαίρι, θα πρέπει να έχουμε ένα κείμενο το οποίο να μην είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο για να μπορέσουμε να δράσουμε άμεσα. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα έχω ένα κατάλογο σκιωδών. Μερικοί είναι παρόντες και άλλοι όχι. Ο κύριος Ανδρουλάκης. Ε, όλοι πιστεύω ότι καλωσορίζουμε την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας Δυστυχώ ο τελευταίο χρόνο αποδείχθηκε ιδιαίτερα θανατηφόρο, αφού πάνω από 100 άνθρωποι πέθαναν στην Πορτογαλία εξαιτία δασικών πυρκαγιών και στην Ελλάδα είχαμε 23 νεκρού από πλημμύρα το μήνα Νοέμβριο. Κανένα κράτο μέλο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τι φυσικέ καταστροφέ τέτοιου μεγέθου. Ε, στο μέλλον, σίγουρα η κλιματική αλλαγή αναμένεται να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο σύνολο και σε άλλε χώρε βέβαια και πρέπει οι εθνικές ε, αρχές να προετοιμάζονται. Σχετικά με το σχέδιο έκθεσης που συζητάμε σήμερα στην Επιτροπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκαρντίνη για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα και να σημειώσω ότι με πολλές από τις τροπολογίες που έχει καταθέσει ε, συμφωνώ στην ουσία. Συγκεκριμένα πιστεύω και εγώ ότι το άρθρο 12 ε, θα πρέπει να αναφέρονται στο άρθρο 12 θα πρέπει να αναφέρονται οι κίνδυνοι για τους οποίους θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και βάσει αυτών να αποφασίζονται οι υλικοτεχνικέ του υποδομές. Ακόμα είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε την επικοινωνία μεταξύ των εθνικών αρχών με την εφαρμογή ενός προγράμματος Εράσμους που αναφέρει και η συγγήτρια καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών ιδιαίτερα με τις χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Στο άρθρο 21 νομίζω ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό τα χρόνια υποχρεωτική συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτική Προστασία να αυξάνονται ανάλογα με το ποσοστό συγχρηματοδότηση. Τέλο, θα ήθελα να εξετάσουμε λίγο παραπάνω το θέμα της διαχείρισης των δυνατοτήτων του Rescue EU. Ε, ο συντονισμό και τελευταίος λόγος πρέπει να ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε περιόδου κρίσεων η διαχείρισή τους θα γίνεται άμεσα και με τρόπο περισσότερο αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ, κυρία Γεντεμάκη. The micro... I think. First, I want to thank the... Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία είναι πολύ κρίσιμη σε τέτοια θέματα προστασία του πολιτή. Όλοι ξέρουμε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα είναι όλο και πιο συχνά στο μέλλον, Μια και προχωράει το θέμα με την άλλαγη του κλίματο. Οι οι πυρκαγιέ, Δυστυχώ θα επηρεάζουν όλο και πιο πολύ το ευρωπαϊκό τοπίο. Επιπλέον, τέτοια περιστατικά θα αυξηθούν σε συχνότητα και φυσικά αυτές οι καταστροφές δεν σταματούν στα σύνορα. Η προστασία του πολίτη είναι στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε από αυτού. Ακόμα όμως και αν συμφωνούμε με την ανάλυση της κατάστασης, υπάρχουν προφανώς ε, διαφορές στο πώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα. Νομίζω ότι το σημείο κίνησης θα πρέπει να είναι η ευθύνη. Πολλοί μου είπαν ότι η βασική αρμοδιότητα, η βασική ευθύνη εξακολουθεί να είναι στις εθνικές ε, αρχές, στα των εθνικών αρχών, στο τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Όλα αυτά λοιπόν καλά και ωραία. Τα κράτη, μέλη και οι αρχές τους ε, είναι άλλωστε και οι πιο κοντινοί φορείς στον πολίτη. Υπάρχει αρχή της επικουρικότητας. Οι εθνικές αρχές είναι οι πλέον αρμόδιες για να αποφασίσουν και να εφαρμόσουν τα προγράμματα διαχείρισης κινδύνου. Θεωρώ ότι είναι προβληματική η μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσουμε τι ικανότητε χρειάζονται. Καταλαβαίνω ότι κάποια κρατημέλη έχουν κάποιες ελλείψεις. Αυτό είναι βασικό πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί η απάντηση να μεταφέρουμε ε, αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρήματα ε, στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Δεν ισχύει έτσι η επικουρικότητα. Επιπλέον, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αντευκρινίζει την αξιολόγηση κινδύνου σε ό,τι αφορά την επιλογή του αντίστοιχου εξοπλισμού. Μπορεί να πρόκειται για εξοπλισμό που έχουν μόνο κάποιες χώρες, αλλά γενικά είναι δύσκολο να υποστηρίξουμε αυτό το γενικό εργαλείο Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητή Πρόεδρε, θέλω λοιπόν να προχωρήσω και να κάνω τι εξή παρατηρήσει. Να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Οι πιο προφανεί εταίροι είναι οι ιονικές χώρε που έχουν τα ίδια προβλήματα, γιατί έχουν το ίδιο περιβάλλον και αυτέ κατά πάσα πιθανότητα θα πλεχθούν από τις ε, καταστροφές και των δεύτερων. Να αναπτυχθεί μηχανισμό προστασία πολίτη χωρίς να έχει αρμοδιότητα τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κατά πόσο θα αναπτυχθούν εθνικές δυνάμει, και θα πρέπει τελικά τον τελικό λόγο να τον έχουν τα κράτη-μέλη. Τρίτον, να βοηθούν τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τα ελλείμματα που έχουν στην ε, στις ικανότητες τους, γιατί η ετοιμότητα είναι μια ολόκληρη νοοτροπία, μια κουλτούρα πρόληψης, πρωτού χτυπήσει η καταστροφή. Όχι τόσο το να στέλνουμε από την Ευρώπη ή από οπουδήποτε εξοπλισμό. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ και έλα. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η ιδέα ενίσχυση μηχανισμών συνεργασία σε θέματα πολιτική προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβάλλεται όταν έχουμε σοβαρές καταστροφές που πλήττουν τις χώρες μας και γειτονικέ χώρες που δεν έχουν και τα απαραίτητα μέσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο κατανοούμε απολύτως. Και βεβαίως σε περίπτωση επιδημίας η συνεργασία είναι πρωταρχικής σημασίας. Σημερίζομαι απόλυτα τις απόψεις της συναδέλφου και βεβαίως πρέπει να πω ότι τα συστήματα πολιτικής προστασίας είναι συστήματα που άπτονται του κάθε εθνικού συστήματος προστασίας. Στη Γαλλία εξαρτώνται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται λοιπόν στα πλαίσια των ε, μεγάλων ε, προβλημάτων, κυρίως ε, με τα θέματα τρομοκρατίας για ένα θέμα το οποίο αφορά όλα τα συναφή εθνικά σώματα ασφαλείας από τους πυροσβέστες, τους ε, αστυνομικούς, σε όλες τις δυνάμεις, το στρατό, το καταλαβαίνουμε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε εκ των προτέρων να είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιου είδους κινδύνους σε επίπεδο κυρίως κρατών. Ε, ώστε να μπορεί να αμήνεται κάθε χώρα και όχι όλα τα θέματα να τα αναθέσουμε στην Κομισιό. Από τεχνικής βεβαίω κοπιάς μπορεί να βοηθήσει η Κομισιό, αλλά πρέπει να πω ότι δεν ε, μπορούμε να δεχθούμε τη μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους για να περάσει το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος και να ευχαριστήσω την Πρόεδρε και την ε, συνάδελφα την κυρία Καρτίνη, για την έκθεση. Νομίζω ότι στο γενικότερο στόχο όλοι συμφωνούμε. Το, οποίο, το μόνο που μας ανησυχεί είναι το πώς το πετύχουμε. Ο στόχο να εισαχθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα για την μετάβαση καταστροφών είναι κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούμε. Όπω είπαν και κάποιοι ομιλητέ όμω, αυτό που είναι σημαντικό είναι στην υλοποίηση να υπάρχει και αναλογικότητα και επικουρικότητα. Εδώ δεν υπάρχει νομική βάση για πλήρη εναρμόρφωσης και είμαι λίγο απογοητευμένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα τόσο σημαντικό θέμα δεν έχει κάνει μελέτη τύπου. Είναι, θεωρώ, αρχή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνεται μελέτη αντικτύπου σε τόσο σημαντικέ δημοφιτικέ προτάσει Εδώ γιατί δεν το έκανε. Τα έπρεπε να το έχει κάνει. Να δούμε τι θα μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν κάνατε μελέτη αντικτύπου. Και για τι ε, τροπολογίε ε, τη κυρία Γκαρντίνη, οι 15 για την ανάγκη τεκμηρίωση. Μπορούμε να έχουμε διαφορετικέ απόψει ε, για την ύπαρξη μη μητρώου, αλλά νομίζω ότι το να αντιβρεθούν αυτέ οι υποχρεώσει και στου ιδιώτε είναι υπερβολικό και αυτό θα δημιουργήσει μόνο περιττή γραφειοκρατία που δεν βλέπω ότι θα εξυπηρετήσει. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η επικουρικότητα. Το είπαν και πολλοί συνάδελφοι σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Εγώ κοιτώντα τη Γερμανία, τι γίνεται με την πυροσβεστική, με τις τεχνικές προδιαγραφές και όλα αυτά, θεωρούμε ότι οι αποφάσεις τελικά θα πρέπει να είναι στα χέρια των κρατών μελών. Και γι' αυτό λοιπόν σίγουρα θα πρέπει να ενισχύσουμε την πτυχή της επικουρικότητας. Σε ένα σημείο υποστηρίζω χωρίς κανένα διχασμό, χωρίς κανένα δισταγμό την ε, εισηγητρία. Το θέμα του εράσμου πώς θα αφαιρεθούν οι πόροι από το εφιστάμενο πρόγραμμα Εράσμου, θα μειωθεί άρα για μια καινούργια, ένα καινούργιο κεφάλαιο. Σίγουρα αποτελεί πολύ επιτυχημένο κεφάλαιο το έράσμου. και θα πρέπει να οργανώσουμε τον τρόπο περαιτέρω χρηματοδότηση και θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και την έλλειψη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι επίκαιρη και καταρχάς καλή. Διότι έχει προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία και αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι να εναρμονίσουμε, διότι δεν, το, δεν πάει προς αυτή την κατεύθυνση η ε, πρόταση, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε και να συντονιστούμε για καταστροφές που ξεπερνούν τη δυνατότητα κάθε κράτους μέλους αν ενεργήσει από μόνο του. Είδαμε τι συνέβη το προηγούμενο καλοκαίρι σε κάποιες χώρες. Γι' αυτό πιστεύω ότι το να μην συμπεριλάβουμε λίστες στις οποίες αναφέρονται οι διάφορες καταστροφές που μπορεί να υποστεί μια χώρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ε, σύγχυση και καταλαβαίνω ότι έχουν ενδιασμού κάποιοι συνάδελφοι, κάποιε πολιτικέ ομάδε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να ενεργούμε λοιπόν από καλού ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι το θετικό και να μην καταλήξουμε σε ένα μηχανισμό ο οποίο κάποια στιγμή θα δούμε ότι δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Μιλώντας για την εν λόγω πρόταση θα ήθελα να σταθώ πρώτα απ' όλα στην πρόληψη. Νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο το θέμα τη πρόληψη. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μία χαρτογράφηση κινδύνων από κάποιες καταστροφές φυσικές στα κράτη-μέλη και να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει ο καθένας να ενεργήσει κάποια συγκεκριμένη στιγμή και να συνεργαστούμε. Πιστεύω ότι δεδομένου ότι έχουμε κάποιες καταστροφές οι οποίες προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, αναγκαστήκαμε κατά κάποιο τρόπο να φτιάξουμε τέτοιου είδους προτάσεις για να τις αντιμετωπίσουμε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσουμε αυτό από την προοπτική την οποία θα έχουμε όταν θα τελειπίσουμε αυτό το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Και κάτι το ειδικό αναφέρεται στο Ταμείο Λιλεγγύη αυτό ο μηχανισμό. Το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε την πρόληψη για να μην συμβεί μια καταστροφή, αλλά τη στιγμή που δυστυχώ κάτι τέτοιο συμβαίνει θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επανορθώσουμε την κατάσταση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε για το Ταμείο αυτό κάποια έκκληση ώστε να είναι το σύστημα αυτό ε, του Ταμείου ε, Αλληλεγγύης βάση κάποιων ε, συντελεστών ε, όπως φερειπίν ο πληθυσμός, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη κάποια προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουν κάποιες πιο αεροκατοικημένες, ε, απομακρυσμένες περιοχές που όντως είναι πιο εκτεθειμένες σε κινδύνους. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ισορροπημένη η πρόταση της Επιτροπής και μιλάμε για έναν μηχανισμό από τον οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε για να καταλήξουμε σε πολύ καλύτερη συνεργασία. Ευχαριστώ. Yes, thank you very much, Chair, and uh, thank you very much. Uh, ο κύριος Φάιτεμα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την κυρία Καρτίνη για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Να τονίσω ευθύ εξ αρχή αυτά που είπε ο κύριο Κίσε και πραγματικά πιστεύω ότι χρειάζεται μελέτη δικτύπου για την πρόταση αυτή. Δεν έγινε. Μετά από πρόταση της Γαλλίας ε, το κοίταξε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή δύο εβδομάδες και μετά κατέθεσε την πρόταση. Ε, λίγο παραπάνω δουλειά μπορούμε να κάνουμε νομίζω. Καταρχά, πιστεύω λοιπόν επίση ότι ο στόχο είναι σαφή. Θα πρέπει να αποτρέψουμε αυτά που είπε ο συναδελφό η σε ό,τι αφορά την ε, σωστή προστασία όταν υπάρχει κάποια καταστροφή. Ο στόχος είναι σαφής, ε, αλλά πιστεύω ότι αυτό αποτελεί και βασικά εθνική αρμοδιότητα. Υπάρχει θέμα και διαφορά μεταξύ ευθύνη και αρμοδιότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μπορεί να βοηθήσει άλλα κράτη-μέλη. Τότε τίθεται θέμα αλληλεγγύης. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται μια σαφή δήλωση αρχικά ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας για να αποτρέψουμε τις ε, καταστροφές. Ύστερα κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γίνεται διαφορά, διαφοροποίηση μεταξύ των κινδύνων ε, ασφάλειας, εθνικές δηλαδή καταστροφές και ε, απειλών ε, ασφάλειας, τρομοκρατία δηλαδή. Υπάρχει λογική και έχει νόημα να γίνεται αυτή η διάκριση, γιατί δεν έχει μεγάλη διαφορά στη τελική ανάλυση από πού προέρχεται ο κίνδυνο. Θα πρέπει να βοηθάμε οι μεν δε. Και ύστερα, η συζήτηση για το κατά πόσον ε, μιλάμε για το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τρίτες χώρες. Εγώ πιστεύω ότι καταρχάς θα πρέπει ένας καλός μηχανισμός για την αρρωγή στο ιστορικό της Ένωσης και για τις τρίτες χώρες να υπάρχει άλλη νομοθεσία. Αυτά λοιπόν ε, για την ε, Ευρωπαϊκό Σώμα Προστασίας του Πολίτη, για το φυσικό δίκτυο και εγώ πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ ότι χρειάζεται μεγαλύτερη άμα, δράση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ομάδα η οποία θα αποστέλλεται στα κράτη-μέλη για να βοηθάει με δικά της ε, μέσα μεταφοράς. Εδώ έχω πρόβλημα γιατί δεν έχει γίνει κυβέρνηση τύπου και δεν υπάρχει και διευκρίνηση για το πώς θα διαμορφωθεί αυτό το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, αν αυτό το Rescue EU ε, έρθει να δράσει στην Ολλανδία, θα έχουν οι Ολλανδικές αρχές ε, αρμοδιότητα και θα μπορούν να αποφασίσουν ή θα αποφασίζει μόνο αυτή η ομάδα, η Rescue U ανεξάρτητα από το που βρίσκεται. Άρα συνολικά χρειαζόμαστε πιο πολλές πληροφορίε και θα πρέπει καταρχά να υπογραμμίσουμε την ε, ευθύνη και την ανάληψη των ευθύνων του καθενός και στην πρόληψη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λίζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την Ελισαβέτα Καρδίνη για τη δουλειά που έκανε. Ομολογώ ότι στους κόλπους του έλεγχα θα πρέπει να το ξεκινήσουμε λίγο, να συζητήσουμε λίγο πιο επισταμένος πρωτού καθορίσουμε τις γραμμές μας. Μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι έγινε με τη μελέτη αντικτύπου, γιατί γίνεται αυτή η πρόταση χωρίς μελέτη αντικτύπου. Όποτε θέλουμε κάτι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολουθούμε μια πολύ αυστηρή διαδικασία. Και εγώ είχα και μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Βέινμαϊρ, ο οποίο μου εξήγησε ότι πάντα χρειάζεται η διαδικασία αυτή της τη και στη συνέχεια αποφασίζει ο κύριο Τίμερμαντς και υπάρχει εντύπωση ότι αν κάποιο έχει διαφορετική άποψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πράγματα κινούνται διαφορετικό. Θα πρέπει να σταματήσει λοιπόν αυτό. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το Κοινοβούλιο. Όταν γίνεται μία πρόταση, θα πρέπει να υπάρχει και μελέτη τύπου. Και ίσως να μην μπορεί να μας μιλήσει για το θέμα αυτό ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά αυτό το μήνυμα θα πρέπει να μεταφερθεί προς τα πάνω στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι δυνατόν να κάνει καθένα του κεφαλιού του, όπως του φαίνεται. Υπάρχουν διαδικασίε. Υποστηρίζω πολλά από τα σημεία τα οποία μας παρουσίασε και μας πρότεινε η Ελίζα Πεταγκαρντίνη σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τον κατάλογο τεχνικών ε, προδιαγραφών που θα πρέπει να είναι λίγο πιο ευέλικτος ο κατάλογος αυτός. Είναι λίγο δύσκολο να αποφανθούμε τι χρειαζόμαστε γιατί δεν χρειαζόμαστε στην παρούσα φάση. Θα πρέπει να αποφασίζουμε λίγο και πρακτικά, επί τόπου. Η αρχή της πρόληψης, πολύ σημαντική. Μπορούμε να την ενισχύσουμε και περαιτέρω. Αν και προσωπικά δεν θεωρώ ότι μπορούμε να εφησυχαστούμε όταν έχουμε ολοκληρώσει την πρόληψη. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι, α, κοιτάξτε, εσείς φταίτε για ό,τι σας συνέβη γιατί δεν φροντίσατε για τη σωστή πρόληψη και την ερώτηση του κυρίου Χάρτεμα. Την έλεγξα για το RESCU. Κατά πόσον ε, αποφασίζει και διατάζει, κατά πόσον αποτελεί ένα προφητικό παράγοντα, ο οποίος εντάσσεται στις δομές των υφιστάμενων εθνικών δομών. Είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό. Είμαι και λίγο διχασμένο για το πώ θα το επιλύσουμε το θέμα, αλλά αυτό που έχω να πω είναι το εξή. Το να πούμε ότι δεν θα κάνουμε τίποτα και θα αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν, ούτε αυτό αποτελεί λύση. Και στις πυρκαγιές στην Πορτογαλία το προηγούμενο έτος, τελικά οι ρωσικές δυνάμεις κατέφτασαν πιο γρήγορα από ότι οι δυνάμεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Και αυτό νομίζω ότι αποτελεί λίγο θέμα για μας. Ε, πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιωθούμε. Ε, τώρα δεν μπορούμε να πούμε και να ισχυριστούμε ότι όλα βαίνουν καλώ και έχουν την ε, ευθύνη του στα μελη Δεν ε, θεωρώ ότι έτσι θα μπορούμε να αρθούμε στο ύψο των περιστάσεων. Τώρα το πώ θα διαμορφωθεί η λύση δεν ξέρω, πρέπει να κάτσουμε να το σκεφτούμε. Και να λεφθούν υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κρατών μελών. Για να καταλήξουμε σε μια πραγματικά καλή λύση. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε κύριε Μάντλ. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την συγγήτρια την κυρία καρτίνη, γιατί ασχολείται πραγματικά επισταμένος με το θέμα αυτό και την ευχαριστούμε. Επί του περιεχομένου, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Πέτερ Λίζα και με αυτά που είπε και ο συνάδελφος Γκίζεκε και ο συνάδελφος Χάιτομα, είναι ξεκάθαρα αυτά που είπαν και θα ήθελα να προστάσω και δύο στοιχεία. Αφενός, μιλάμε για μια κεντρική διαμορφώση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τις δυνάμεις που χρησιμοποιούνται ε, στο πλαίσιο. Αλλά αυτές οι δυνάμεις θα πρέπει να είναι τοπικές ή περιφερειακές ε, και θα πρέπει να ακολουθείται η επικουρικότητα, την οποία και υπογράμμισε ιδιαίτερο η κυρία Καρτίνη. σα ευχαριστώ πολύ. Θεωρούμε λοιπόν ότι η αρχή τη επικουρικότητα εδώ θα πρέπει να τονιστεί. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να στραφούμε σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του ΡΕΣΚΙΓΙΟΥ. Προβλέπεται την οργάνωση ευρωπαϊκού διαγωνισμού για την ε, χρήση των μέσων. Και σε χώρες ε, που αναφέρθηκαν πυρκαγιές στην Ιταλία αλλά και σε άλλα μέρη στην Ευρώπη όπου υπάρχει σύστημα προστασίας από καταστροφές το οποίο βασίζεται βασικά σε εθελοντές. Εδώ θέλουμε να προειδοποιήσουμε και να αποτρέψουμε ενδεχόμενη εμπαραγματοποίηση του κλάδου αυτού της προστασίας από καταστροφές. Αυτό πραγματικά θα το επέκρινε διδέρως υπογραμμίζω ιδιαίτερα τα θέματα συγχρηματοδότησης και για μέσα τα οποία δεν έρχονται από τον κορβανά αυτό. Και ενδεχομένω ε, να πρέπει να αναφερθούν και ρητά οι κίνδυνοι και να αναφερθούμε και να κοιτάξουμε το θέμα της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Φαίνεται πως όχι. Ο Διευθυντής Λούχνερ έχει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της. Είναι πολύ χρήσιμη και νομίζω ότι εισακούστηκε και η άποψη του Συμβουλίου. Θα ε, επισημάνω τα σχόλια και θα σταθώ σε αυτά. Αλλά καταρχήν κινούμαστε με βάση την επικουρικότητα όπως διέπεται από το άρθρο 196. Όποια και να είναι η λύση θα πρέπει να εξευρεθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο και αυτό κάνουμε σε αυτή την πρόταση. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να κινηθεί περαιτέρω αλλά δεν κινήθηκε λόγω επικουρικότητας. Ε, σε σχέση με την προετοιμασία και την ανταπόκριση. Ως προς τη μελέτη αντικτύπου θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω και να πω ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε θεσμικά ζητήματα. Μπορώ να σας πω όμως πώς ανέκυψε αυτή η πρόταση. Είχαμε μία ε, ευρωπαϊκή μελέτη αποτίμησης κινδύνου όπου συνεισέφεραν όλα τα κράτη-μέλη και έναν ορισμό των χασμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη πριν από τις καλοκαιρινές ε, πυρκαγιές. Ορίσαμε τα χάσματα, ιδιαίτερα σε σχέση με τα καταφύγια, της ε, δασικές πυρκαγιές πυρκαγιές και ούτω καθεξής. Το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή του μας είπε ότι μπορούμε να απλουστεύσουμε το πλαίσιο λειτουργίας και είχαμε και μία εξωτερική ανεξάρτητη αξιολόγηση. Και του χρόνου θα υποβάλουμε μία νέα πρόταση. Γνωρίσαμε και τις καλοκαιρινές ε, πυρκαγιές και θα ήθελα να πω ότι Πρόκειται για μια πολύ ευρία ε, έννοια και χρονική ε, στιγμή γιατί άρχισε από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Εμείς θεωρούμε ότι αρχίζει τον Ιούνιο και λίγη τον Σεπτέμβριο. Είχαμε 200 νεκρούς, 100 εκ των οποίων από την Πορτογαλία. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ερεύνησε το ζήτημα και του είπαμε τον Οκτώβριο ότι προσπαθήσαμε να κινητοποιήσουμε μέσα αλλά δεν τα βρήκαμε και δεν τα βρήκαμε έγκαιρα. Άρα ο Πρόεδρος θεώρησε ότι το ζήτημα είναι επίγον γιατί χρειαζόμαστε επίγουσα δράση αν δεν θέλουμε να έχουμε και άλλους ε, νεκρούς και οικονομική ζημία, γιατί το θέμα πραγματικά έχει επίγοντα χαρακτήρα. Αν δείτε την πρόταση, καταρχήν εστιάζει την προσοχή της στα κράτη-μέλη, στα ε, πάγια στοιχεία ενεργητικού των κρατών μελών που συγχρηματοδοτούν με την Επιτροπή. Και αυτό που έχει σημασία είναι η εθελούσια βάση στοιχείων ενεργητικού. που διαθέτουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να συγχρηματοδοτήσει σε υψηλότερο ποσοστό, διότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη βοήθεια μεταξύ κρατών μελών. Γιατί συμφωνούμε ότι πρόκειται για πρωταρχική ευθύνη των κρατών μελών. Με αυτή τη σειρά έχετε την τοπική, περιφερειακή και κρατική ανταπόκριση μετά τη διμερή βοήθεια και μετά την κοινή βάση. Και μετά έχετε στοιχεία ε, ενεργητικού RESC-EU. Ε, Η νομοθεσία τέθηκε σε εφαρμογή το 2013 και σε 30 περιστάσεις τα κράτη-μέλη δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, δηλαδή δεν βρήκαμε τα μέσα για να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν ξεκίνησε πέρσι το θέμα δηλαδή. Πέρσι ήταν ε, πολύ σοβαρές οι συνέπειες βέβαια. Το θέμα της επικουρικότητας να το λάβετε υπόψη γιατί δεν έχουμε ούτε την ε, δυνατότητα ούτε και την φιλοδοξία να προβούμε σε άμεση πολιτική προστασία στα κράτη-μέλη. Ζητούμε μία λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά. Πέρυσι, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, υπήρχαν αυτά τα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επειδή ο καθένας αντιμετώπιζε υψηλό κίνδυνο, δεν υπήρξε επιμερισμός. Εάν λοιπόν δεν λειτουργεί αυτό το κρατικό σύστημα, θα πρέπει να έχουμε πάγια στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι στις Βρυξέλλες, αλλά στα κράτη που βρίσκονται κοντά στον κίνδυνο. Και μόνο όταν και εάν ένα κράτος μέλος ε, προβάλλει μία ε, ε, αίτηση, τα μέσα αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Άρα παίρνουμε μία στρατηγική απόφαση. Όλες ε, οι ε, επιχειρησιακές λύσεις ε, γίνονται σε επίπεδο κρατών μελών. Βεβαίως το επιχειρησιακό παραμένει σε επίπεδο κρατών μελών και κρατικών αρχών και η Επιτροπή παίρνει μια στρατηγική απόφαση χρήσης μέσων. Δηλαδή ακόμα και να θέλαμε δεν θα, μπορέσουμε, δεν θα μπορούσαμε να αναλάβουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Ως προς το Εράσμους έχουμε ένα πρόγραμμα ε, ανταλλαγών που χρηματοδοτείται από, την, ε, από τον προϋπολογισμό πολιτικής ε, προστασίας αλλά η ανταλλαγή αυτή γίνεται μέσα σε μερικές μέρες ή δύο εβδομάδες το πολύ. Θα έπρεπε να επεκτείνουμε αυτό το διάστημα. Συμπερασματικά, εμείς είμαστε μία επιχειρησιακή δύναμη. Ε, έχουμε να λάβουμε αποφάσεις τάχιστα μέσα σε 24 ώρες. Αυτό είναι ε, δύσκολο όταν υπάρχει μια περίπλοκη νομική βάση και επειδή το δικαστήριο μας είπε ότι υπάρχουν περιθώρια απλούστευσης, προσπαθήσαμε να απλουστεύσουμε τους δείκτες ε, συγχρηματοδότησης. Ο λόγος για τον οποίο αποκλείσαμε στην ε, πρόταση συγχρηματοδότηση εκτός της κοινή βάσης ήταν ο λόγος που ανέφερε και η εισηγήτρια. Δεν ξέρουμε τι μέσα υπάρχουν. Εξαρτόμαστε από τα κράτη-μέλη και αν δεν έχουμε μία προσφορά από κράτη-μέλη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρετε αν θα λάβετε απάντηση ως κράτος μέλος από άλλα κράτη-μέλη με βάση το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών πολιτικής προστασίας. Άρα αποζητούνται άλλες λύσεις. Γι' αυτό και πέρσι είχαμε τρίτες χώρες που βοήθησαν τα κράτη-μέλη σε πολλές περιστάσεις γιατί έδρασαν τάχιστα. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ποια είναι τα μέσα για να είμαστε λειτουργικοί και γρήγοροι. Οποιαδήποτε πρόταση αυξήσει την ευελιξία μας, για μας θα ήταν ευπρόσδεκτη. Τέλος, πέρα από το γεγονός ότι εστιάζουμε την προσοχή στα κράτη-μέλη και την εθνική κυριαρχία, κατά, την, ε, κατά το αίτημα βοήθειας, εάν υπάρχει επιχειρησιακός έλεγχος, ε, τονίζουμε τη σημασία της πρόληψης και της ε, προετοιμασίας. Και αυτό γιατί βασιζόμαστε στο άρθρο 196 αλλά είπαμε ότι θα δούμε πώς μπορούμε και αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαρθρωτικά, τα διαρθρωτικά ταμεία ε, με βάση τις κλιματικές αλλαγές και την ε, πρόληψη. Ε, έχουμε επαφή με τους συναδέλφους από τις γενικές, ε, γενικές διευθύνσεις γεωργίας, κλίματος και περιβάλλοντος έτσι ώστε να υπάρχουν να πληρούνται αυτοί οι όροι της προετοιμασίας. Η κυρία Γκαρντίνη, για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και την Επιτροπή που νομίζω ότι απάντησε διεξοδικά στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν και που σχετίζονται και με τη δική μου έκθεση Είμαι πεπισμένη ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή εργασία. Αυτή η εργασία θα ξεκινήσει, ξεκίνησε από την προηγούμενη φοιτεία, με βάση την αρχή της επικουρικότητας, γι' αυτό και μίλησα για την ενίσχυση του συστήματος ως προς συμμετοχή των περιφερειακών και εθνικών αρχών, γιατί αυτό, αυτός είναι και ο πολικός αστέρας που μας ε, καθοδήγησε μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας. Αυτό το οικοδόμημα δεν θα το θίξουμε. Θα κινηθούμε μέσα στα πλαίσια του με βάση την αρχή της επικουρικότητας, διότι η πολιτική προστασία δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Η πολιτική προστασία είναι κάτι που προέρχεται από τις περιφέρειες. Δηλαδή στη χώρα μου που δυστυχώς έχουμε μεγάλη πείρα, η πρώτη υπεύθυνη είναι η δήμαρχη. Και από εκεί ανεβαίνουμε τις κλίμακες. Δηλαδή όταν δεν τα καταφέρνει ο Δήμαρχος τότε απευθύνεται στην περιφέρεια και μετά στις κρατικές αρχές. Αλλά πέρσι είχαμε βοήθεια και από το Μαρόκο γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε τα δικά μας αεροσκάφη. Άρα, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν επιφυλάξεις, στην πραγματικότητα συμβαδίζουμε με την ε, προσέγγιση που θέλουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι με τη συνεισφορά όλων θα ορίσουμε καλύτερα αυτές τις καταστάσεις έτσι ώστε να ερμηνευθούν σωστά και να κινηθούν προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε. Υπενθυμίζω ένα στοιχείο που υπενθυμίζω πάντα. Υπάρχει το ευρωβαρόμετρο το οποίο είναι σταθερό. Το 90% των Ευρωπαίων ε, πολιτών ε, τάσεται υπέρ της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας και θέλει να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση όταν οι κρατικές αρχές δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Να χτυπήσουμε ξύλο αλλά με τις ε, τρομοκρατικές ε, ενέργειες που ζήσαμε και επειδή μπορούν να επανεμφανιστούν, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο, ελπίζοντας ότι δεν θα συμβεί ποτέ. Αλλά στην προηγούμενη θητεία είχαμε θελήσει να εντάξουμε αυτό το κεφάλαιο. Θα μιλήσουμε για ε, ιδιαίτερα περίπλοκα μέσα, οπότε δεν μπορούμε να ζητήσουμε τη σύνδρομη 27 κρατών μελών. Θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή βάση και ελπίζω ότι θα προωθήσουμε μια καλή βάση για τους ε, πολίτες και αυτό το είδαμε και από τις πρόσφατες ε, δημοσκοπήσεις, γιατί η ασφάλεια είναι το πρώτο μέλημα των πολιτών μας και θα πρέπει να φανεί ότι δρούμε άμεσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγη. Πληρώνεται η συζήτηση επί αυτού του θέματος. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 10 Απριλίου στις 11 το πρωί και προβλέπεται ψηφοφορία στην ΕΜΒΗ 16-17 Μαΐου. Περνούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχουμε στη ημερήσια που έχουμε. Η χρηστή διαχείριση των ε, φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες, η περίπτωση των δασών. Ε, έχει ζητηθεί σχέδιο γνωμοδότησης και θα μας το παρουσιάσει η συντάκτρια γνωμοδότηση, κυρία Κονέτσκα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι τιμή μου που μπορώ να σας παρουσιάσω το κείμενο αυτό. Μιλάμε για τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες υπέρ του Ισοδασών. Και είναι πολύ φατικό το γεγονός ότι ζητήθηκε γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ότι στη τελική ανάλυση αυτό άμα σχετίζεται ασφαλώς με την επίτευξη των βιώσιμων στόχων. Είναι δύσκολο το θέμα. Αλλά είναι σημαντικό να αρχίσουμε καιρός, γιατί η προστασία των δασών είναι απολύτως απαραίτητη, ιδιαίτερα των ε, παρθένων δασών και είμαι πεπισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ έχει υποχρεώσεις έναντι των τρίτων χωρών. Κατανοούμε το γεγονό ότι όλα τα κράτη-μέλη θέλουν να αναπτυχθούν περαιτέρω και ότι αυξάνεται ο πληθυσμό του. Προφανώ λοιπόν είναι δύσκολο να επιληθούν τέτοια προβλήματα και χρειάζονται περίπλοκα μοντέλα. Και έτσι λοιπόν να μην, χωρίς να βλάπτονται το περιβάλλον. Και χαίρομαι που συμφωνεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρόβλημα όμως είναι διαφορετικό. Την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή α, μας παρουσίασε μία έκθεση για την αποδάσωση και χαίρομαι που επιτέλους δημοσιεύτηκε. χρειάζεται για ένα καλό σχέδιο δράση. και γι' αυτό λοιπόν προκύπτει ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αποδάσωση και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και αυτή να αποτελεί ε, μέλος της λύσης, μέρος της λύσης του προβλήματος. Αυτό έχει να κάνει και με την ε, τήρηση των δεσμεύσεων που αναλάβουμε στο Παρίσι. Χαίρομαι λοιπόν για τις τροπολογίες που λάβαμε και τις οποίες θα κοιτάξουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Ελπίζω λοιπόν θα καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία, όπως και στην πρόταση για την αναδιαμόρφωση των δασών. Σημαντικό είναι να αγωνιστούμε μαζί, γιατί το πρόβλημα κατά βάση δεν είναι πολιτικό. Το θέμα είναι οι επόμενες γενιές να μπορέσουν και αυτές να επιζήσουν και να ζήσουν σε ένα κατάλληλο περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, πρόεδρο Πρόεδρος. Ισκαιώτης, οι συγητές, μόνο η κυρία Πετήρ βλέπω να είναι παρούσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, πρόεδρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και προφανώς ε, ως ΕΛΚΑ θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες, αλλά να πω δύο λόγια για το θέμα αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το γεγονό τη αλλαγή του κλίματο είναι κάτι το αδιαφεσβήτητο, το ζούμε κάθε μέρα. Καθημερινέ είναι ειδήσει για βία και απρόβλεπτα μετεωρολογικά φαινόμενα. Η Κροατία έχει πληχθεί ιδιαίτερω ε, πρόσφατα. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν πολιτικέ οι οποίε θα εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας περισσότερο από ότι 1,5 βαθμό μέχρι τα τέλη του αιώνα, όπως και δεσμευτήκαμε στο Παρίσι. Αλλά πολύ απλά δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο και θα πρέπει πλέον να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας. Να βοηθήσουμε λοιπόν τις αναπτυσσόμενες χώρες να συνεργαστούν μαζί μας. Η ευθύνη για τη διαχείριση των δασών είναι μια σημαντική πτυχή. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία θα στέσει τα σωστά κριτήρια, τις ε, σωστές πολιτικές για να πετύχουμε την μείωση της αποψήλωσης. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε όμως ότι και οι πολιτικές μας θα μειώσουν τις δασικές εκτάσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει να προσμετρούνται λοιπόν τα αποτελέσματα και το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να φροντίσουμε να μην επιβαρύνει απλά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους παραγωγούς, Απαγορεύοντα ουσιαστικά την πρόσβαση στις αγορέ, ε, το οποίο και συνέβαινε έως τώρα. Οι Κροάτε ε, κατασκευαστές ε, επιπλοποί διαμαρτύρονται, γιατί σε κάποια τμήματα του κόσμου, όπως για παράδειγμα στην Ινδία, στην Βόρεια Αφρική, αντιμετωπίζουν εμπόδια. Και αυτό ως αντίπεινα στα δικά μας εμπόδια τα οποία την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέλει να εφαρμόσει τους ευρωπαϊκούς ε, κανόνες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το φροντίσουμε. Και δυστυχώ διαπιστώνω ότι στις πιο πολλές περιπτώσεις ε, αυτοί που πλήττονται είναι η μικροπαραγωγή στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λεκή Πρόεδρος. Άλλος, κανείς το θέμα αυτό. Όχι. να στραφώ προς την κυρία Μέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι όντως τα βάση είναι μέρος της ε, πλούσιας φύσης και αποδίδουν ε, κέρδη, ωφέλη κοινωνικά και άλλα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά για την πλανήτη, για την ειρήνη, για την ευημερία των πολιτών. Και ξεπερνούν βεβαίως τα εθνικά σύνορα. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα αγαθό παγκόσμιο και πρωταρχική σημασία. Όπως ξέρετε, το θεματολόγιο της αηφόρου ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, έχει μιλήσει για τη σημασία της αηφόρου εκμετάλλευσης των δαθών, πράγμα που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε καλύτερη διακυβέρνηση. Όντως, η διαφάνεια και η αξιοπιστία είναι πρωταρχική σημασίας ώστε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα δάση σφαιρικά και ιδίω στα πλαίσια της αυξημένης πίεσης που υφίστανται. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την συνεργασία της δικής σας Επιτροπής για την γνωμοδότηση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πολύτιμο αυτό το οποίο κάνατε για τα δάση και τι αναμένετε να γίνει για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τα ωφέλη της πολιτικής μας στα πλαίσια της ε, δράσης FLEX και του προγράμματός μας. Το πρόγραμμα FLEX φέτος γιορτάζει την 15η επέτειό του και είναι συνεργασία μεταξύ ε, κρατών, μελών, τρίτων χολών, ε, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα κατά της ε, αρνητικής και παράνομης εκμετάλλευσης των πόρων των δασών μας έχουν συναυθεί ε, γύρω στις 15 εταιρικές συμφωνίες με τρίτες χώρες και Έχουμε την υποστήριξη των ιδιωτικών φορέων και γενικότερα την ε, κοινοτήτων των διαφόρων στα όλα στις χώρες μας και στις τρίτες χώρες και εδώ έχουμε και την περίφημη ε, συμφωνία περιξηλίας η οποία διέπει την ε, συμφωνία αυτή. Προσπάθειες λοιπόν εκ όλων Πρόβλημα να βελτιώσουμε την κατάσταση και το επενθυμίζω. Όπως αναφέρθηκε πολύ σωστά από την εισηγήτριά σας, πέραν της παράνομης ε, ξύλωσης υπάρχουν και άλλες απειλές για τα δάση. Από την επέκταση της ε, γεωργίας, ε, από την εκμετάλλευση των γεών, από την εκμετάλλευση των διαφόρων καλλιεργειών και η αποψήλωση των δασών επίσης είναι ένα πολύπλοκο θέμα που δημιουργείται σε πολλές χώρες από τη σύμπραξη διαφόρων συντελεστών. Ελπίζουμε ότι την Παρασκευή η δημοσίευση δύο μελετών θα βοηθήσει την ε, ανάπτυξη της ε, δικής σας γνωμοδότησης. Οι μελέτες έγιναν από ανεξάρτητους συμβούλες. Η μία αφορά την μελλοντική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποψήλωση των δασών και η δεύτερη αφορά τις, ε, αντικ, τους αντικτύπους, ε, τις περιβαλλοντικούς και άλλους, τις ε, The της παραγωγής και χρησιμοποίησης του φινικελαίου. Ε, οι μελέτες αυτές είναι πολύ σημαντικές ελπίζω και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πρέπει να αποφασίσουν ποια είναι η πορεία που θα ακολουθήσουν για την προστασία των δασών στο μέλλον. Ευχαριστούμε. κυρία Κόνετσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Προς την Επιτροπή. Είμαι πεπισμένη ότι οι αποφάσεις σας ε, δεν θα χρειαστούν τόσο πολύ μεγάλο χρόνο όσο χρειάστηκαν οι μελέτες για να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι η απόφαση που θα πάρουμε συγκεκριμένα για το φινικέλ. Η πολιτική αποψήλωση των δασών δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Τουλάχιστον εγώ δεν τα βλέπω έτσι τα πράγματα και την γνωμοδότησή μου δεν την έκανα με αυτό το πνεύμα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο αφορά το μέλλον όλων. Και είμαι πεπισμένη ότι με τους συναδέλφους, τους συνεισηγητές θα βρούμε μια κοινή γλώσσα ώστε το μέλλον των δασών να είναι όσο πράσινο όσο θέλουμε να είναι και τα ίδια μας τα δάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται και η συζήτηση από αυτού του θέματος. Τροπολογία κατάσταση τροπολογιών 22 Μαρτίου 11 το πρωί. Συζήτηση και ψηφοφορία το Μάιο. Το επόμενο θέμα είναι το μέλλον των τροφίμων και τη γεωργίας. Σχέδιο γνωμοδότησης για την άγκρη. Σύμφωνα με το κανόνα 53.1, η κυρία Ωζελίκ Ντολαέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι, όντως πρόκειται για μια γνωμοδότηση που αφορά το μέλλον της ΚΑΠ και των ειδών διατροφής. Είναι θέματα τα οποία παρακολουθούμε στην Άγκρη του Σύνεγγες. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, διότι η πολιτική αυτή είναι μία από τις ιδρυτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες γενικές θετικές παρατηρήσεις όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ αυστηρό. Η τελευταία μεταρρύθμιση του 2013 δεν έχει τεθεί σε ισχύ σε κάποιες χώρες και βλέπουμε πάλι να επανέρχεται το θέμα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι χρειαστήκαμε 13 μήνες για να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση για την ε, μήνυ μεταρρύθμιση που ονομάστηκε Omnibus. Εάν μας αποστέλει λοιπόν στο τέλος Μαΐου η Κομισιόν την, Επιτροπή, την πρότασή της, θα έχουμε μόνο 9 μήνες να επεξεργαστούμε το θέμα αυτό και θα είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Υπάρχουν και τα ερωτηματικά ε, του προϋπολογισμού καθώς και τα συμπεράσματα τα οποία ακολουθούν από το Brexit. Καταλαβαίνετε ότι θίθεται και θέμα διαδικασίας. Θα έπρεπε να περιμένει τα αποτελέσματα της έκθεσης πρωτοβουλίας της Επιτροπής Άγκρη από τον κύριο Νότφερ για να συμπεριλάβει στην πρότασή της και τις θέσεις που θα εκφραστούν εκεί. Βλέπω λοιπόν δύσκολα πώς μπορούμε αν πάρουμε όλο αυτό το θέμα στα χέρια μας τέλος Μαΐου να προχωρήσουμε ε, που θα μπορούσαμε να τα ψηφίσουμε όλα αυτά τον Ιούνιο. Μας ασκεί λοιπόν μεγάλη πίεση η Κομισιό. Δεν μπορούμε παρά να προχωρήσουμε με στρατιωτικό βήμα. Γι' αυτό χρειάστηκε εγώ την έκθεσή μου τη συντάξω αγγλικά που δεν είναι η μητρική μου γλώσσα το ίδιο συμβαίνει και με τις τροπολογίες. Και αυτό είναι πραγματικά λυπηρό για μία μεταρρύθμιση σε έναν τομέα που είναι ιδιαίτερη σημασία. Έτσι εκτίθεται η Επιτροπή στον κίνδυνο να γίνει πολύ βιαστικά η δουλειά μας. Εάν εξάλλου δεν, γίνει, ε, δεν υιοθετηθεί το κείμενο πριν από το Μάιο 2019 δεν θα υπάρχει καμία δέσμευση για τους διαδόχους μας και την επόμενη Επιτροπή επί της ουσίας του άλλου θέματος. Επί της ουσίας τώρα. Έχουμε, ε, όπως καταλαβαίνετε, να κάνουμε με ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα τόσο της γεωργίας και όσο του περιβάλλοντος. Προτείνω λοιπόν αυτά τα δύο θέματα να τα εξετάσουμε από κοινού. Η πολιτική η τομεακή θα πρέπει να ε, οδηγήσει τους, οδηγούς, τους ε, γεωργούς να οδηγούνται σε καλύτερες πρακτικές και να μπορέσουν να προχωρήσουν προς την επίτευξη δύο στόχων στη γεωργία και στον σεβασμό του περιβάλλοντος. έχουμε λοιπόν δύο πυλώνες. Στον πρώτο πυλώνα έχουμε τις άμεσες βοηθείες που χορηγούνται μετά από αυστηρές περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Στο δεύτερο πυλώνα στρεφόμεθα στην στρατηγική την τομεαθή και της περιοχής, αλλά που με τη δημιουργία κινήτρων, για να μπορέσουμε να έχουμε επενδύσεις έρευνα και καινοτομία σε τοπικό επίπεδο. Η ιδέα ενός τρίτου πυλώνα που αφορά μέτρα διαχείρισης κρίσεων είναι κάτι που επίσης θα πρέπει να μελετήσουμε. Η ΚΑΠ θα πρέπει επίσης να έχει μια πραγματική προσδοκία και φιλοδοξία προς τις νέες πράσινες πηγές ενέργειας και θα αναφέρω και ως παράδειγμα και την δημιουργία φυτικών πρωτεϊνών μεταξύ άλλων. Όσον αφορά τι εμπορικέ συμφωνίε, θα πρέπει η ΚΑΠ να εγγυάται ότι κάθε είδο διατροφή και κάθε αγροτικό ε, προϊόν ανταποκρίνεται στι ίδιε απαιτήσει στον υγειονομικό, στον κοινωνικό, στον περιβαλλοντικό τομέα, όπω όλα τα άλλα ε, ευρωπαϊκά προϊόντα. Εγώ επειδή ε, κάνουμε γνωμοδότηση, χρειάστηκε να περιοριστώ σε μία σελίδα για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο ενδιαφέρον και με μεγάλη ενδιαφέρον, αναμένω τις αντιδράσεις σας συνάδελφοι, ξέρουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών έχει οριστεί για την επόμενη εβδομάδα 27 Μαρτίου στις 11 το πρωί. Ευχαριστώ. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ποιος θα ήθελε το λόγο. Ο κύριος Εκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άξιοι συνάδελφοι. Σε διάφορα άρθρα της Ευρωπαϊκής Συνθήκης ε, στο 3.9.168 αναφέρεται ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, ως σκοπό να προαγάγουν την ευημερία των λαών και ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασία. Και έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι οι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκρίνονται και να συνάδουν με τη στοχοθεσία τη συνθήκη και να δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στην υγεία των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε θέματα κοινωνική ισότητα και σε θέματα προστασία του περιβάλλοντο. Γιατί όλοι είμαστε θύματα των φυσικών καταστροφών, αλλά σε πολλέ αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχω την εντύπωση ότι αυτέ οι προτεραιότητε συχνά ε, δεν λαμβάνονται σημαντικά υπόψη για το 20% του προπολογισμού 2014 έως 2020 για προστασία των, ε, του κλίματος και στα σχετικά μέτρα. Αλλά οι πόροι αυτοί τελικά πού καταλήγουν. Και εκτιμάται ότι οι αξιολογήσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το προσύνισμα τη ευρωπαϊκή πολιτική ε, ε, αγροτική πολιτική είναι πάρα πολύ υπερβολικά αισιόδοξε. Άρα πολλά έχουμε να κάνουμε ακόμα σε ό,τι αφορά το 70% ε, των εκπομπών του του άνθρακα που προέρχονται από την παραγωγή του κρέατος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τι σημαίνει η μείωση της βιολογικής παραγωγής στην Ευρώπη, πράγμα το γεγονός ότι η παραγωγή και η κατανάλωση ζωικών προϊόντων αναφέρεται συχνά ότι θα πρέπει να μειωθεί και αυτό θα οδηγούσε σε πρασινίσμα της πολιτικής, αλλά παρόλα αυτά δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. Θα πρέπει να εστιαστούμε πολύ περισσότερο στην υγεία όλων των πολιτών και στην ποιότητα ζωής αλλά και στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ζώων. Γιατί αυτό έχει άμεσες θετικέ επιπτώσεις ε, και για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον. Μόνο τα εμπορικά συμφέροντα των επιχειρήσεων δεν μπορούν να κυριαρχήσουν ε, και να καθοδηγούν τις αποφάσεις μας, γιατί αυτό δεν ανταποκρίνεται στο συμφέρον του, των πολλών. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να καταστήσουμε την γεωργία ως κινητήριο δύναμη της οικονομίας και χρειαζόμαστε λοιπόν όλα τα στοιχεία αυτά. Θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει με όλα αυτά τα σκάνδαλα με τα τρόφιμα. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, μπορούμε να λάβουμε ρόλο προστασίας ε, του περιβάλλοντος και των ζώων. Θα πρέπει η νέα ΚΑΠ να εξασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων μας, να είναι καλύτερη σε όλο τον κόσμο. Αλλά δυστυχώ στην γνωμοδότηση αυτή δεν αναφέρονται τα σημαντικά αυτά θέματα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ε, υπογραμμίζονται επαρκώς. Και αφού του διάβασα, λοιπόν, ε, την ε, έκθεση της συναδέλφου μου, φάνηκε, λες, και διαβάζαμε μία έκθεση της Επιτροπής Άγκρη ή των ενώσεων των χρετών. Δεν είδα σκληρή κριτική για το σύστημα αυτό το οποίο έχει οδηγήσει σε τόσα πολλά υπαρξιακά προβλήματα πολλές επιχειρήσεις και για να συνοψίσουμε. Αν δεν ε, τι θα σέψουμε αυτή τη βιομηχανική αγροτική παραγωγή θα μας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και γι' αυτό λοιπόν θα καταθέσω τροπολογίες για την καλύτερη ευημερία και προστασία των ζώων, πιο πολύ προστασία των ζώων, πιο πολλά μέσα για ασφαλή ε, και υγιεινή παραγωγή τροφίμων, πιο πολλά μέσα για την τοπική παραγωγή, βιοπικιλότητα, προστασία αυτή, σε μεγαλύτερη προστασία για τις ε, οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μείωση των πόρων για που ασχολούνται με την εντατική καλλιέργεια και εκτροφή ζώων. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ, Λεκύπρο. Ευχαριστώ, Λεκύπρο. Κανείς άλλος. Η ε, κυρία Μελιόρθα, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την κυρία Τελαέ για την έκθεση της. Συμφωνώ με τις ανησυχίες ό,τι αφορά την προθεσμία. Σε λίγο θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες ορόσημο για την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση. Αν έχουμε την γνωμότησή μας και μετά την έκθεση της Επιτροπής ε, Γεωργικών Υποθέσεων, κάπως θα δυσκολευτούμε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφορετική σειρά σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση. Εν πάση περιπτώσει τώρα δεν αλλάζουν τα πράγματα, αλλά ανησυχώ και εγώ όπως είπατε. Δεύτερο σημείο. Και εγώ πιστεύω ότι η Γεωργία στο μέλλον θα πρέπει να συνεισφέρει πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης. Σε κάποια σημεία συμφωνώ και με τον Προλαλήσαντα. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν πιο επισταμένως. Πώς θα μπουν σε μια τόσο μικρή γραμματότηση δεν γίνεται. Επίσης, με ανησυχεί και το εξή. Η βιώσιμη γεωργία συχνά αντιμετωπίζεται ω συνάρτηση του μεγέθους της επιχείρησης. Εμείς πιστεύουμε ότι όσο πιο μικρή ε, μάλλον υπάρχει η εντύπωση ότι όσο πιο μικρή είναι η επιχείρηση, αν είναι οικογενειακή, τόσο πιο καθαρά εργάζεται, τόσο πιο πολύ προστατεύει το περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό εφάπαξ. Ε, θα πρέπει να κοιτάμε σε κάθε περίπτωση πόσο βιώσιμη είναι μια επιχείρηση, πώς θα πετύχουμε την επιστηστική ασφάλεια, πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα αυτά. Και δεν νομίζω ότι όλα εξαρτώνται πια από το μέγεθος της επιχείρησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η πρόεδρο. Άλλο κανεί. Μάλιστα. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον κύριο Ανιώτη. Can, can someone help him? Μπορεί κάποιος να τον βοηθήσει. Ή να μετακινηθείτε. Yes, very well. Τώρα με ακούτε, εντάξει. Επιλύσαμε το τεχνικό ζήτημα. Θα ήθελα να σχολιάσω την παρούσα κατάσταση. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τη διαδικασία, διότι εξαρτάται από δύο άγνωστους παράγοντες, το μέγεθος των ΜΜΕ μετά το Brexit και την κατάσταση δεν μπορούμε να τη διασαφηνίσουμε τώρα. Και γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να τονίσω τα τέσσερα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από την ανακοίνωση της Επιτροπής. Με βάση τα σχόλια, τα δικά σας σχόλια. Με την ανακοίνωση η Επιτροπή θέλει να έχει μία ε, μεγαλύτερη περιβαλλοντική ε, αντιμετώπιση της ΚΑΠ και να συνδυάσουμε το οικονομικό και περιβαλλοντικό σκέλος της ΚΑΠ. Ένα από τα πιο θετικά στοιχεία που έχουμε μετά από τις δημόσιες ε, διαβουλεύσεις για την προετοιμασία της ανακοίνωσης που είδαμε όταν προετοιμάσαμε την μελέτη αντικτύπου είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου με τις νέες τεχνολογίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την οικονομική και την ε, περιβαλλοντική απόδοση με βάση συνέργειες τη στιγμή που το σύστημα παροχής συμβουλών θα λάβει υπόψη τις τεχνολογίες εχμής. Επίσης θα πρέπει να έχουμε καλύτερη στοχοθέτηση υποστήριξης. Αυτό δεν έχει να κάνει με το μέγεθος. Το μέγεθος είναι ουδέτερο. Αυτό που μετράει είναι οι δυνατότητες διαχείρισης αλλά ο τρόπος ε, κατανομής ε, του χρήματος είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο θα ενταχθεί στην επικουρικότητα. Επίσης, να βασιζόμαστε περισσότερο στη γνώση και σύνδεσμα μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και συμβουλευτικών συστημάτων και τέταρτο στοιχείο καλύτερη ισορροπία μεταξύ σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών μελών και δικαιούχων με στόχο να μετακυλήσουμε αυτές τις πολιτικές από τους ελέγχους στην αποδοτικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν έλεγχοι στο μέλλον, ούτε ότι δεν ελέγχουμε την αποδοτικότητα, αλλά θα υπάρξει αυτή η μετακίνηση προς καλύτερη αποδοτικότητα. Επίσης, όπως προείπατε, ε, μας απασχολούν και ζητήματα υγείας μέσα στα πλαίσια της ΚΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη το μυς, όπως τον έλεγχο των αντιβιωτικών που δεν έχει σχέση μόνο με τα ζώα αλλά και με τους ανθρώπους. Και επίσης καλύτερο προσανατολισμό της πολιτικής έτσι ώστε οι γεωργοί να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανησυχίες των καταναλωτών. Τέλος, ως προς τη διαδικασία υπάρχει ένας πλούτος πληροφοριών που είναι διαθέσιμος σε σχέση με τη νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ λαμβάνοντας υπόψη την ε, ε, τεκμηρίωση που υπάρχει για τη μελέτη αντικτύπου. Κάτι το οποίο συνοψίστηκε σε μία δημόσια διάσκεψη για να γνωρίζει το κοινό καλύτερα για το τι πιστεύουμε ε, για την πολιτική αυτή πριν περάσουμε στις νέες προτάσεις. Ευχαριστούμε πολύ η κυρία Ντελάη για να συνοψίσει. Ευχαριστώ πρόεδρε εντάχει. Ανταποκρινόμενοι σε αυτά που είπαν συνάδελφοι, όπως ο κύριος Εκ, θα ήθελα να εμβαθύνω ορισμένα ζητήματα, αλλά σε οκτώ μέρες ε, δεν είναι εύκολο να συντάξει κανείς μία γνωμοδότηση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε πολύ περισσότερα. Σε σχέση με αυτά που μας είπε ο κύριος Ανιώτης, νομίζω ότι μας ενδιαφέρει η διπλή αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων και η μετάβασή τους προς αυτή τη διπλή αποδοτικότητα. Έλαβε υπόψη τα σχόλια των συναδέλφων και θα βασιστώ στις δικές σας προτάσεις τροπολογιών για να ολοκληρώσω αυτή τη γνωμοδότηση η οποία θα πρέπει να ψηφιστεί πολύ σύντομα. Τουλάχιστον οι τροπολογίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 27 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγη η συζήτηση επί του θέματος αυτού. Το επόμενο θέμα Και για να συμπληρώσω, συγγνώμη και εγώ, θα ήθελα να πω ότι θα ψηφίσουμε στην ΕΜΒΗ στις 25-26 Απριλίου και η τροπολογία είναι μόνο στα Αγγλίκα. Το επόμενο θέμα είναι μία ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερόμενους ε, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις πλαστικές ύλες, αλλά επειδή έχουν αρχίσει, αργήσει οι ενδιαφερόμενοι και επειδή προβλεπόταν η συζήτηση στις 4.30 θα πρέπει να περιμένουμε την ώρα εκείνη για να προβούμε στην ανταλλαγή απόψεων με τους εμπειρογνώμονες. Άρα διακόπτουμε μέχρι τις 4.30.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 Hello, Σας καλωσορίζω στην ε, ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερόμενους για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Πλαστικές Ύλες. Ε, το οργανώνουμε με βάση την ε, πρωτοβουλία, ίδια πρωτοβουλία για την στρατηγική για τα πλαστικά και αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της κυκλικής ε, ε, οικονομίας. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους ενδιαφερόμενους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να σας μιλήσω για αυτούς. Η κυρία Σάσκια Βάλρεντ που είναι ε, ε, σύμβουλος για την βιώσιμη ανάπτυξη της Εσένσια που ασχολείται με χημικά, Emma Prisland, η οποία ασχολείται με τους θαλάσσιους ρήπους και τις θάλασσες υποκίνδυνο, η κυρία ε, Πατρίσια Βανκελούβε που είναι διευθύντρια του, των, ε, των καταναλωτών και των υποθέσεων περιβάλλοντος στο Plastics Europe και η κυρία ε, Άρο Ματιλά, η οποία ασχολείται με στα πλαίσια της εταιρείας Atria Plastics με την ε, ε, συσκευασία. Και ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο κύριος Σαντάουσκας. Ο πρώτος ομιλητής έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου. Το ναι, άναψε το μικρόφωνο. Ναι, να κάνω λοιπόν την εισαγωγή μου, αλλά θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Μια και δεν έχουμε και χρόνο στη διάθεσή μα και βασικά αυτό που μα απασχολεί είναι θέλουμε να ακούσουμε του εμπειρογνώμονε. Και θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε, γι' αυτό και καλέσαμε τόσο πολλού εμπειρογνώμονε. Να σα καλωσορίσουμε λοιπόν στην Επιτροπή μα. Σα ευχαριστώ ιδιαίτερω γιατί ήταν ε, ε, πολύ πρόσφατη η πρόσκληση. Το πλαστικό είναι ένα υλικό με το οποίο φαίνεται ότι το αντιμετωπίζουμε ε, πολύ με μεγάλη σπατάλη και χάνουμε πολλά. Χάνουμε πολλά για το περιβάλλον, για την οικονομία. Η πρόκληση σαφώς είναι να αντιμετωπίσουμε το πλαστικό με βιώσιμο τρόπο στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Ε, και θα καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό αν όλοι οι φορείς ε, κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Και θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτή. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονό ότι μπορεί να γίνει ανταλλαγή απόψεων με τι εμπειρογνώμονε και προσβλέπω στο συναρπαστικό αυτό το δίχω άλλο απόγευμα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρο, και τώρα να δώσω το λόγο στου ε, προκεκλημένου μα. Ε. Ο κύριος Πέκης Βαντάν Μπάρμπετ. Η κυρία μάλλον. Ναι, αν θα μπορούσα να... Η κυρία Βάλρετ, αν θα μπορούσα να έχω και την παρουσίαση. Κατά σας ευχαριστώ που μας καλέσατε. Για την παρουσίαση λοιπόν της κυρίας Βάλρετ. Σα ευχαριστώ που μας καλέσατε λοιπόν σε αυτή την επιτροπή και θα θέλαμε να κάνουμε μία σύντομη παρουσίαση τη ΕΣΕΝΣΗ. Η Βαλκική Ομοσπονδία τη της Χημικών και και ανθρώπινων επιστημών έχουμε μια ξεχωριστό τμήμα σε ό,τι αφορά την παραγωγή τέτοιων ε, προϊόντων, την Essential, την οποία και εκπροσωπώ εδώ, σε ό,τι αφορά την στρατηγική για τα πλαστικά. Καλωσορίζουμε ορίζουμε την ε, στρατηγική για το πλαστικό, η οποία θα δημιουργήσει μια νέα νοοτροπία και θα μας οδηγήσει σε καινούργια επιτεύγματα, θεωρούμε. Διαπιστώνουμε με μεγάλη μας χαρά ότι αναγνωρίζεται φυσικά η αξία των ε, συμφετικών υλικών στην πολιτική αυτή για το πλαστικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και όντω ε, τα συμφετικά υλικά δεν ε, μπορούμε να τα θεωρήσουμε απλά ως απορρίμματα. Είναι πολύ πιο πολύτιμα. Είναι τμήματα της κυκλικής οικονομίας σε ό,τι αφορά τους πόρους στην Ευρώπη, τη δημιουργία της εργασία, την καινοτομία. Τρία ζητήματα που μας απασχολούν ιδιαίτερα στην εσένσια. πιστώνουμε λοιπόν ότι επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στις ε, συσκευασίες ε, πλαστικού, όπου σε πολλές περιπτώσεις στη δημοσιότητα προωθείται η ιδέα ότι ό,τι είναι πλαστικό, ό,τι είναι συμφετικό αποτελεί πρόβλημα. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Καταρχάς, να... ένας από τους στόχους μας είναι να αυξήσουμε ε, το ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών στις συσκευασίες. Κοιτώντας λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία βλέπουμε ότι ανακυκλώνται στην παρούσα φάση 40% του πλαστικού μόνο. Και αυτό είναι από όρια διάφορων επιλογών που έχουν γίνει ήδη σε ό,τι αφορά την ευθύνη, για παράδειγμα, του παραγωγού, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα τα οποία εστιάζονται σε υλικά όπως το PET και HDPE τα οποία δεν ανακυκλώνονται ιδιαίτερω ή σχεδόν καθόλου. Και όχι επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωση των υλικών. Όλα τα θερμοπλαστικά πολυμερή ουσιαστικά μπορούν να περάσουν από μηχανική ανακύκλωση. Αυτό έχει να κάνει μαζικά από τι επιλογέ που γίνονται και από το γεγονό ότι πάντα σήμερα οι γραμμικέ επιλογέ είναι πολύ εύκολε και πολύ φθηνέ. Για παράδειγμα, πολύ συχνά καταλήγουν σε χωματερές εκτός Ευρώπης αυτά τα πλαστικά απορρίμματα και πιστεύουμε ότι σημαντική ευθύνη φέρνει και η ίδια, φέρει και η ίδια η βιομηχανία σε ό,τι αφορά τις συσκευασίε, για παράδειγμα. Εξακολουθούμε να μην δίνουμε επαρκή σημασία σε ένα σχεδιασμό για την κυκλικότητα Και ο οικολογικό σχεδιασμό σίγουρα λοιπόν αποτελεί μια λύση. Πιστεύουμε επίση ότι η απαγόρευση τη Κίνα, China Ban, το γεγονό ότι δεν ε, επιτρέπονται και κάποια υλικά στην Κίνα θεωρούμε ότι δεν είναι πρόβλημα ιδιαίτερο, αλλά αποτελεί μια ευκαιρία. Ευκαιρία να κρατήσουμε τα υλικά μα εδώ στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι θα πρέπει να υπάρξει η επένδυση σε τοπικέ και περιφερειακές μονάδες ανακύκλωση και θα πρέπει φυσικά να υπάρχει επαρκή κλίμακα επαρκείς ικανότητες και καταστάσεις για την ανακύκλωση των προϊόντων και κυρίως να υπάρχει ανακύκλωση και για κάποια είδη πολυμερών. Είναι λοιπόν σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό κλίμα επενδύσεων για το μέλλον. Επίσης, αναφέρεται και το ποσοστό ανακυκλωμένου περιεχομένου για κάποια θέματα, για κάποια προϊόντα σε τα πλαίσια των πράσινων δημοσίων συμβάσεων. Είναι σημαντικό καταρχάς να ορίσουμε έναν σαφή ορισμό. Τι εννοείται με το ποσοστό ανακυκλωμένου περιεχομένου. Τι συνυπολογίζεται. Επίσης, θα θέλαμε να κάνουμε το εξής σχόλιο. Το ποσοστό θα επικεντρωθεί στην ποσότητα. Εμείς δεν θέλουμε μόνο ποσότητα, θέλουμε και ποιότητα υλικών, των ανακυκλωμένων υλικών. Και για να πετύχουμε λοιπόν την ποιότητα των ανακυκλωμένων υλικών θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα πιστοποιητικό, ένα σύστημα πιστοποίηση για όλη την Ευρώπη πρωτού καταστεί υποχρεωτική η ανακύκλωση συγκεκριμένη ποσότητα ε, υλικών. Τέλος, ε, θα θέλαμε να πούμε ότι η ανακύκλωση, ε, πέρα από την ανακύκλωση πρώτη γενιά δεν είναι απαραίτητα μόνο downcycling. Σε κάποιες περιπτώσεις εφόσον πρόκειται για παιδική ανακύκλωση. Το θέμα της ανακύκλωσης δεν αποτελεί πρόβλημα. Το θέμα της ε, μεθόδου ανακύκλωσης, το οποίο ε, και της μεθοδολογίας ανακύκλωσης, σίγουρα αποτελεί μια λύση. Η, πλαστική, η στρατηγία του πλαστικού θα επιδραθεί επίσης σε θέματα καινοτομία. Είναι σημαντική φυσικά η καινοτομία και ως Ευρωπαίοι και Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Χημικών και Πλαστικών εδώ έχουμε να δραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη μηχανική ανακύκλωση, που και πάλι θα πρέπει να εντάξουμε συγκεκριμένες ουσίες ε, επιτάχυνσης κτλ. Αλλά σε ό,τι αφορά και τις καινοτομίες για τη χημική ανακύκλωση, γιατί αυτό θεωρούμε ότι δεν τονίζεται παρκώς στη στρατηγική για, την πλαστική, για τα πλαστικά. Και θεωρούμε ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική εναλλακτική και θα πρέπει να αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποσότητα υποχρεωτικής ανακύκλωσης, γιατί αποτελεί μία λύση για υλικά, όχι τόσο πολύ για συσκευασίε, αλλά για άλλες χρήσεις και αποτελεί και μία λύση η οποία θα αφαιρούσε τα πιο επιζήμια συστηκτικά από το πλαστικό. Τέλος, η βιομηχανία συμμετέχει ιδιαίτερως για την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, όπως για παράδειγμα τη χρήση του διεξιδίου άνθρακα ως πόρο και θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμο όλα αυτά. Έχουμε διάφορα πολιτικά προγράμματα και έχουμε και την ανάπτυξη εναλλακτικών ζωοτροφών θεωρούμε ότι αυτό θα αποτελεί μια λύση που θα έχει και οικονομικά ωφέλη και οικολογικά ωφέλη σε ό,τι αφορά τη χρήση εναλλακτικών πόρων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα απορρίμματα και τα λύματα. διαπιστώνουμε ότι είναι στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής, αλλά δεν υπάρχει ουσιαστικά δημόσια ευθύνη. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Πρόκειται για μια κοινή ευθύνη όλων μας. σε ό,τι αφορά και το κοινό, αλλά και τις αρχές. Είναι λοιπόν αρμοδιότητα των δημοσίων αρχών. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι αποποιείται την ευθύνη τη η βιομηχανία. Πιστεύουμε ότι η βιομηχανία θα πρέπει να ακολουθήσει μια θετική προσέγγιση ε, προληπτικά, όπως για παράδειγμα με, το, με την άσκηση Clean Sweep με το λιμένα της Αμβέρσας και τους παραγωγούς πολυμερών και τον τομέα της επιμελητίας συμφωνήθηκε να υπάρξει πρόληψη της ε, μόλυνσης αυτής και επενδύουμε ιδιαίτερως και σε κατάρτιση και εκπαίδευση και βλέπετε λοιπόν ε, το πλάστη μομπίλ αυτό το φορτηγό στην φωτογραφία κάτω, όπου Έχουμε το ειδικό αυτό, του ειδικού οι οποίοι πάνε από σχολείο σε σχολείο και ενημερώνουν τα παιδιά για το πώ γίνεται η ανακύκλωση και πραγματικά το πιστεύουμε ότι έχει μεγάλη επιτυχία αυτό το πρόγραμμα. Τέλο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ανακοινωθεί και κάποιε εθελούσιε δεσμεύσει σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση τη στρατηγική για την αύξηση τη ε, ανακύκλωση, προκειμένου να αποφύγουμε τελικά τα υλικά αυτά να καταλήγουν ω σκουπίδια στο περιβάλλον. Επίσης, έχουμε και δράσεις ενέργειες σε ό,τι αφορά τις ε, άσκησεις καθαρισμού του λιμένου της Αμβέρσιας, αλλά και άλλες τέτοιες, ε, άλλα εγχειρήματα σε ό,τι αφορά τα μικροπλαστικά και τις ε, σχετικές προτάσεις. Πεστιφεύουμε ότι θα πρέπει να περιορίζεται σε μικροπλαστικά τα οποία έχουν προσθεθεί σκόπιμα. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου να μην καταλήγουν στη φύση. Είναι σημαντικό τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται να είναι προφανώς αναλογικά και να υπάρχει και σαφής ορισμός του τι ακριβώς εννοείται και τι ρυθμιστικές ε, επιλογές υπάρχουν, όχι μόνο στο πλαίσιο αυτό, αλλά να εξετάζεται και κατά πόσο μπορεί να αποφευθεί ε, κίνδυνος, ε, ο κίνδυνος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πλαστικά για την ε, μία και μοναδική χρήση, διαπιστώνουμε ότι λείπει ορισμό του τι είναι τελικά το single use plastics και θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί, αν θέλετε, και παράδοξο γιατί τα πλαστικά δεν είναι από τη τους. Δεν προορίζονται για μία και μόνο χρήση και το γεγονός ότι τα θεωρούμε ε, ως υλικά για μία χρήση, σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία. Και επικεντρωνόμενοι σε αυτά τα πλαστικά μία χρήσεως, δεν θεωρώ ότι μπορούμε να καταφέρουμε την αλλαγή της νοοτροπία και της κουλτούρας που επικρατεί στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να περάσουμε στην ε, όλο και πιο περιορισμένη χρήση των ε, υλικών μίας χρήσης, γιατί θέλουμε προφανώς να κολυμπάμε σε θάλασσες χωρίς ε, σκουπίδια. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση των ε, πλαστικών. Αυτά είναι λοιπόν ε, επιγραμματικά τα ζητήματα που μας απασχολούν. Ξέρω ότι τα είπα γρήγορα γρήγορα, αλλά αν έχετε ερωτήσεις ευχαριστώ να τις απαντήσω. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα η κυρία Πρίσλαντ έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Good afternoon. Thank you very Καλό σας απόγευμα. Είμαστε μία ευρεία μη κυβερνητική και είμαστε υπέρ της ε, ε, συμμαχίας ε, πλαστικών και ζητάμε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι ελεύθερο από πλαστικές ύλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει κατανοήσει πολύ καλά. Η, οικονομική, ευρωπαϊκή οικονομία βασίζεται στο ε, πλαστικό το οποίο δεν στοιχίζει έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία αλυσίδα. Το 40% χρησιμοποιείται για τη συσκευασία και πολύ μεγάλο μέρος αυτού δεν ανακυκλώνεται. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η συσκευασία αυτή οδηγεί, η συσκευασία αυτή οδηγεί σε μείωση ε, λιμάτων ε, τροφίμων. Αλλά η λογική μας είναι ότι έτσι έχουμε μάθει με την ταχύφαγία και πολλές φορές μας πείθουν ότι το εμφιαλωμένο νερό είναι καλύτερο από το νερό της βρύσης, αλλά έτσι παράγουμε περισσότερα πλαστικά από αυτά που μπορούμε να διαχειριστούμε. Όταν ανακυκλώνουμε ένα μικρό μέρος ε, στα σύνορά μας και ε, εξάγουμε το υπόλοιπο ή το θάβουμε, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά με το σύστημά μας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει δραστική μείωση και η κυκλική οικονομία να γίνει πραγματικότητα, καθώς και να έχουμε καλύτερη διαχείριση των πλαστικών που χρησιμοποιούμε. Αυτό θα πρέπει να υποβοηθηθεί από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όταν μιλάμε για συνολική μείωση χρήσης πλαστικού, τι σημαίνει. Θα πρέπει να μην χρησιμοποιούμε επιβλαβή πλαστικά. Καλωσορίζουμε την ε, Επιτροπή η οποία μιλά για μικροπλαστικές ύλες και ε, οξοδιασπάσιμες, κάτι το οποίο θα ήταν πολύ σκοπιμότερο. Ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε τα επιβλαβή αυτά προϊόντα να μην χρησιμοποιούνται πλέον στην αγορά. Επίσης, η στρατηγική οδηγεί σε άλλες ε, πηγές ε, μικροπλαστικών όπως το πέλετ θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ρυθμιστική ε, πρόταση όπως ισχύει με τον κανονισμό περί ξυλίας. Η εθελούσια ε, προσέγγιση δεν ε, οδηγεί σε πραγματικό έλεγχο και αυτό δεν είναι επαρκές για τις μικροπλαστικές ύλες. Άρα για να μειώσουμε τη χρήση πλαστικών θα πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση πλαστικών υλών μίας χρήσης. Η νομοθετική πρόταση της Κομισιόν είναι πολύ σημαντική για τη μείωση της ε, ρήπανσης από πλαστικά. Και αυτό το βλέπουμε στις ε, παραλίες κυρίως. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα αίτια και να αποτελέσουμε παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα σε όλες μας παραλίες έχουμε γόπες, ε, συγκεκριμένα συσκευασίες, ακόμα και καλαμάκια, πλαστικά ποτήρια και ούτω καθεξής. Για να είναι αποτελεσματική αυτή η νομοθεσία θα πρέπει να οδηγήσει σε συλλογή στοιχείων. Για να δούμε ποια στοιχεία είναι στην αγορά. Υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία ως προς αυτό για να έχουμε ε, μία ιδέα θεωρούμε ότι θα πρέπει να ποσοστοποιήσουμε τα στοιχεία αυτή. Δείχνουμε ότι 46 δις πλαστικά ε, ποτήρια χρησιμοποιούνται, 16 εκατομμύρια φλιτζάνια, μάλλον ε, ποτήρια για καφέ και επίσης ε, ε, συγκεκριμένα ε, προϊόντα take-away τα οποία ανέρχονται σε 2,5 δις. Θα θέλαμε να έχουμε μείωση στους στόχους που να μπορούν να επιτευχθούν μέσω συγκεκριμένης φορολόγησης και τελών. Αυτό θα οδηγήσει σε πιο σωστή χρήση πλαστικού. Θα σταματήσω για να μιλάω για τα πλαστικά μίας χρήσης, αλλά υπάρχουν και άλλες ε, πλαστικές ύλες. Θα πρέπει να έχουμε ε, μία δασμολόγηση και επιβολή τελών για τις πλαστικές ύλες. Θα πρέπει να έχουμε ένα νέο σχηματισμό και προγραμματισμό έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη χρήση αυτών των προϊόντων, δηλαδή νέα χρήση. Και αυτές οι πλαστικές ύλες αφορούν και ύλες συσκευασία που μπορούν να αναβαθμιστούν και να έχουν ανακύκλωση 100%. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη η Εάν χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό θα πρέπει να είναι ασφαλές για τους ανθρώπους και για το περιβάλλον. Αν δεν υπάρχει όμως ε, ανιχνευσιμότητα δεν θα, έχουμε, ε, δεν θα μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα δευτερογενή πλαστικά. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι προσθετικές χημικές ουσίες επίσης είναι επιβλαβείς και ίσως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καν. Και τέλος, ε, για να έχουμε μία καλύτερη εικόνα, δεν θα πρέπει να έχουμε ε, ψευδολύσεις γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά τα αναλώσιμα και ανακυκλώσιμα δεν αποτελούν ε, ασφαλή λύση για το περιβάλλον. Χρειάζεται ρύθμιση και εποπτεία αυτών των υλικών, καθώς και καλύτερη σήμανση για το πώς θα πρέπει να απομακρύνονται. Ε, θεωρώ ότι τα πλαστικά που βασίζονται σε βιοηλικά θα πρέπει να έχουν, ε, να λάβουν υπόψη ότι δεν μπορούν να έχουν χρήση στη θάλασσα. Υπάρχουν πολλά υλικά που γράφουν με κεφαλαία «δεν είμαι πλαστικό», αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για το πώς θα πρέπει να απομακρυνθούν. Πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη διαχείριση των πλαστικών για την προώθηση της ανακύκλωσης θα πρέπει να υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει επαναχρησιμοποίηση όπως ορίζει και η οδηγία περί συσκευασιών και αυτό αφορά και την ανακύκλωση με βάση μία ιεράρχηση. Μέσα στα πλαίσια της ανακύκλωσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος. Επίσης, πώς γίνεται η συλλογή των πλαστικών. Εμείς ως Συμμαχία είμαστε υπέρ της στρατηγικής πλαστικών και περιμένουμε τα νέα μέτρα τα οποία θα προταθούν. Τα πιο επίγοντα είναι η νομοθεσία για τα πλαστικά μίας χρήσης τα οποία θα πρέπει να ενταχθούν στην οδηγία γιατί οι υπεύθυνε βιομηχανίες έχουν αυτές, αυτά τα στοιχεία. Επίσης η στρατηγική θα πρέπει να βελτιωθεί ως προς την ε, μεταχείριση των πλαστικών και επαναχρησιμοποίηση. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 800.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει μία αίτηση για τη μείωση της χρήσης των πλαστικών και αυτό διευρωπαϊκά. Άρα θα ήθελα να σας ζητήσω ως Επιτροπή να αποστείλετε ένα σαφές μήνυμα προς την εκλογική σας βάση, έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο σωστή προσέγγιση για τη χρήση των πλαστικών. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Βάγγελουβε έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ πέρα να σας κάνω την παρουσίαση αυτή και η παρουσίαση αυτή θα γίνει στα αγγλικά σε ό,τι αφορά το, το ε, ε, εκπροσωπώ. Είμαστε μια πανευρωπαϊκή οργάνωση ανά την Ευρώπη με έδρα στις Βρυξέλλες και εκπροσωπούμε πάρα πολλές ε, κατασκευαστές καθώς και ε, κατασκευαστές πλαστικών συσκευαστιών και άτομα τα οποία ασχολούνται με την ε, μετατροπή, με την μεταποίηση των πλαστικών. Ε, σε επίπεδο απασχόλησης έχουμε περισσότερο από 1,5 εκατομμύρια άτομα, εταιρείες περισσότερες από 60.000, περισσότερες μιμιέ, ε, κύκλο εργασιών 350 δις και στην καινοτομία είμαστε από τους καλύτερους. Θα ήθελα να μιλήσω πρώτα απ' όλα για την αύξηση της συνειδητοποίησης της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης που είναι κάτι πολύ σημαντικό σε όλη τη ζωή κάτι προϊόντος, από την αρχή ως το τέλος. Και θα πρέπει για να αρχίσουμε αυτή την επαναχρησιμοποίηση, να αρχίσουμε από την ε, συλλογή, την των ε, ε, διαφόρων συσκευασιών και πλαστικών υλών που θέλουμε να ε, ανακυκλώσουμε. Επίσης, ο οικολογικός σχεδιασμός των πλαστικών υλών είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι ένας από τους στόχους της κυκλικής οικονομίας, ώστε να έχουμε στη, ε, πόρους αποδοτικούς και ε, σε πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπή διοξιδίου του άνθρωπος. Επίσης, είναι σημαντικό να δούμε πώς θα κάνουμε τον σχεδιασμό των προϊόντων που θα έχουν ε, οικολογικό σχεδιασμό. Αυτοί οι οποίοι διαθέτουν τα εμπορικά σήματα είναι αυτοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί και θα πρέπει να είναι οι απαιτήσει περισσότερο προς την ποιότητα παρά προς την ποιότητα. Τα στάνταρ, οι κανόνες θα πρέπει να γίνονται ε, σεβαστή και θα πρέπει όλοι να αναλάβουν σε θελούσια βάση δεσμεύσεις για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη χρήση και ανακύκλωση. Ένα ε, πολύ σημαντικό και δεύτερο στοιχείο της στρατηγικής σας είναι πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μη λιγότερες ε, λιγότερα απορρίμματα, λιγότερα απόβλητα. Να δούμε πρώτα απ' όλα τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε λιγότερα ε, απόβλητα, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τη συλλογή, να, την, ε, τα συλλέξουμε, να κάνουμε τη διαλογή, να τα ναι, ε, να χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, η ευαισθητοποίηση Τη συμπεριφορά των ατόμων είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει όλοι να ξέρουν ότι ένα προϊόν το οποίο θέλουν να χρησιμοποιηθεί πρέπει να συλλέγεται, να γίνει τη διαλογή του και στους κατάλληλους χώρους για να μπορέσει να επαναχρησιμοποιηθεί. Επίσης, θα πρέπει, όπως σας είπα, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος της ζωής αυτών των προϊόντων. Υπάρχει πρόβλημα με τα απορρίμματα, μπορούμε να κάνουμε έναν διαφορετικό σχεδιασμό. Και θα ήθελα εδώ να κάνω κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις. Όταν μιλάμε για πλαστικές ύλες μίας χρήσης, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δώσουμε ένα σωστό ορισμό. Πρόκειται για την χρήση κυρίως του προϊόντος και βεβαίως ε, πρέπει να επικεντρωθούμε στο υλικό που χρησιμοποιείται για να μειώσουμε ε, την ε, χρήση τους, την εμφάνισή τους παντού, στους κάδους απορριμμάτων, στις παραλίες. Και βεβαίω, δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοιους ε, απαγορεύσει που να οδηγούν τον καθένα να ρίχνει το πρόβλημα στην πλάτη του αλουνού. Επίσης, Ξέρουμε ότι στον τομέα της καινοτομίας μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε ε, για την κυκλική οικονομία να συσχεριστούμε αυτό το θέμα της καινονομίας. Η κύκλος ζωής των πλαστικών προϊόντων, η χρησιμοποίησή τους και το ότι θα χρησιμοποιούμε νέες ε, πηγές ενεργειακές και δεν θα ε, εξαρτώμεθα από τις παραδοσιακές ε, πηγές ενέργειας και από τα ορικά κάψιμα είναι κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε βελτίωση της κατάστασης. Θα πρέπει επίσης να έχουμε προϊόντα με πλαστική ύλη τα οποία μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε, να μεταποιήσουμε και βεβαίως πώς θα δώσουμε περισσότερη ζωή στο τέλος της ζωής ενός προϊόντων και πώς θα μπορέσουμε να τα ξαναεπαναχρησιμοποιήσουμε. Και βεβαίως ο οικολογικός σχεδιασμός είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικός. Επίσης, ε, θα πρέπει για να γίνεται καλύτερα η ανακύκλωση να προστίθενται ε, διάφορες ύλες μέσα στα πλαστικά που χρησιμοποιούμε ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερο καιρό και πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τη διαλογή πιο εύκολο. Χαιρετίζουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική και έχουμε να μοιραστούμε κοινού στόχους. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε ως Plastics Europe την, ε, μια δημοψήφιση την οποία ονομάζουμε η εθελούσια δέσμευσης για τα πλαστικά του 2030. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το επιτύχουμε μέσω δραστηριοτήτων ε, που θα ε, κάνουμε πάρα πολύ ε, προσβάσιμη σε όλους. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε την έκκληση πλαστικών στο περιβάλλον. Πώς θα μπορέσουμε να ε, μειώσουμε το ότι διάφορες παλέτες φόρτωσης, εκφόρτωσης προϊόντων χάνονται ή χρησιμοποιούνται μια φορά. Πώς θα κάνουμε την ε, μέτρηση των ε, ε, διαφόρων το, τον, ε, του κύκλου ζωής των διαφόρων προϊόντων για να μπορέσουμε να τα ε, ξαναχρησιμοποιήσουμε. Και όπως σας είπα, επαναλαμβάνω ότι ο οικολογικός σχεδιασμός είναι πολύ σημαντικός. Και το τι κάνουμε στο τέλος της ζωής των πλαστικών και πώς τα επαναχρησιμοποιούμε είναι κάτι που επίσης θα μας βοηθήσει. Η Plastics Europe είναι ε, μια εταιρεία η οποία θέλει να ασχοληθεί με τα θέματα της έκκλησης των πλαστικών και τα απόβλητα και τα απορρίμματα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε για θέματα που αφορούν λύσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον περισσότερο από 355 σχέδια σε 40 χώρες. Και επίσης για... συνεργαζόμαστε στα πλαίσια πρωτοβουλειών με το Παγκόσμιο Συμβούλιο περί πλαστικών στα πλαίσια προώθησης ε, και συνεργασίας προτάσεων στα πλαίσια της UNEP καθώς και του G7 και του G20. Ε, είναι πάρα πολύ επί, παρα, ε, ε φιλόδοξοι στόχη μας, μόνο έτσι πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε καλά αποτελέσματα. Επίσης θέλουμε να υπάρχει δέσμευση την οποία θα αναλάβουν ε, διάφοροι φορείς εκτός και εντός της βιομηχανίας των πλαστικών. Να ε, επιταχύνουμε την καινοτομία για τον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων και το 2040 να φτάσουμε σε 100% επαναχρησιμοποίηση κυρίως 60% χρησιμοποίηση της συσκευασίας πλαστικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ο μιλητής είναι ο κ. Μάκη Μαδηλά. Έχετε το λόγο. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μας για την ε, πολύ σημαντική αυτή η ευκαιρία να παρουσιάσουμε και εμεί ε, την απόψή μας ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά στην κυκλική οικονομία. ονομάζομαι Άρωμα Κιμάτλα και ε, εκπροσωπώ την Άτρια, μια μεγάλη ε, φιλανδική εταιρεία τροφίμων. Σκοπός μας είναι να παράγουμε βιώσιμα και περιβαλλοντικά υπεύθυνα ασφαλή τρόφιμα. Επίσης θέλουμε να ε, συνδραμούμε στην δημιουργία πιο ασφαλών και πιο βιώσιμων συσκευασιών. Για να συνοψίσουμε, αυτά είναι τα βασικά έξι θέματα τα οποία πρέπει να είναι στον πυρήνα τη συζήτησή μα, θεωρούμε. Η ασφάλεια τροφίμων πάντα θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Αυτό το λέω και το τονίζω. Οποιαδήποτε νέα εξέλιξη και ανακάλυψη και εφεύρεση θα πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό αυτό. Η πρόληψη είναι καλύτερος τρόπος για την ε, διαχείριση των απορριμμάτων και άλλα μέτρα φυσικά είναι πολύ σημαντικά. Αλλά να υπογραμμίσω ότι μόνο η ανακύκλωση δεν ε, μπορεί να μας εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα. Οι καλύτερες συσκευασίε λοιπόν ε, μειώνουν την σπατάλη τροφίμων. Η σπατάλη τροφίμων είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τη νέα ε, συσκευασία. Και γι' αυτό λοιπόν η συσκευασία πάντα θα πρέπει να προοδεύει το προϊόν και να περιορίζει κατά συνέπεια την σπατάλη τροφίμων. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι διαπραγματεύσεων. Η δημιουργία αξία ε, είναι ένα βασικό φορέα για την βιωσιμότητα. Τι μάθαμε λοιπόν, ότι η πρόοδο μπορεί να επιτευχθεί μόνον όταν υπάρχει προτίμηση από πλευρά του καταναλωτή ή ό,τι καλή δουλειά και να κάνουμε μπορεί να πάει χαμένη. Επικεντρωνόμαστε επίσης σε, μια ολιστική συνολική προσέγγιση. Ο καταναλωτή αντικτύπωση για το περιβάλλον θα πρέπει να είναι ο οδηγό μας. Σε κάθε βήμα τη Αλυσίδα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα τον αντίκτυπο που υπάρχει στο περιβάλλον. Η μόλυνση με σκουπίδια αντιμετωπίσετε με τον καλύτερο τρόπο με προγράμματα, με επικοινωνία με τον καταναλωτή. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν σωστή συλλογή και επικοινωνία με τον καταναλωτή. Βλέπετε λοιπόν τον οδηγό που ακολουθήσαμε την τελευταία δεκαετία. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο και για το μέλλον. Ο λόγος είναι ότι είδαμε πόσο πρακτικά αποτελέσματα είχε αυτός ο οδηγός. Και το καλύτερο παράδειγμα ήταν η νέα πρωτοποριακή συσκευασία για το κύμα που ξεκίνησε το 2017. Φανταστείτε να υπήρχε παρόμοια προσέγγιση σε ευρία κλίμακα Σκέφτεται τι γίνεται στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας που πηγαίνετε. Τις δυνατότητε ε, περιορισμού του πλαστικού που υπάρχουν. Τι καταφέραμε λοιπόν να κάνουμε. Μείωση πλαστικού που χρησιμοποιείται κατά 50% για ένα προϊόν. Σήμερα, 12 μήνες μετά από την εισαγωγή του προϊόντος αυτού, διαπιστώνουμε ότι οι καταναλωτές τέτοιου είδους εξέλιξης θέλουν ε, και απαιτούν να γίνουν σε άλλες κατηγορίες προϊόντων. Και αυτό είναι προφανώς ε, επειδή είναι τόσο εύκολο να γίνει εμφανής ε, η διαφορά. Και όλα αυτά φυσικά στην ε, μικρή κλίμακα της Φιλανδίας, αλλά 50% πραγματικά είναι μεγάλο ποσοστό. Ο βασικός λόγος που πήρε το βραβείο αυτό το προϊόν είναι ότι αύξησε την αποτελεσματικότητα του υλικού σε ό,τι αφορά την ανάλυση που έγινε για τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Η μείωση του αποτυπώματος ήταν, του άνθρακα ήταν πιο πολύ από 30% και όλοι οι δείκτες σε ό,τι αφορά την παραγωγή, την ε, κατανάλωση ενέργειας, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και όλα αυτά η νέα συσκευασία δεν είναι τέλεια από πλευρά ανακύκλωση, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια τεράστια πρόοδο. Ένα μεγάλο βήμα προ την βιωσιμότητα των συσκευασιών. Η πρόοδος λοιπόν σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα θα πρέπει να θεωρηθεί σε συνάρτηση και με άλλες βελτιώσεις. Δηλαδή οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη στην αξία ή στην αξία όπως γίνεται αντιληπτή, θα ανέκοπτε αυτές τις θετικέ εξέλιξεις. Ο ρόλος λοιπόν της συσκευασία είναι τελικά να προστατεύσει την, ε, το τρόφιμο. Άρα οποιαδήποτε επιδείνωση της προστασίας του, τροφίμου θα έχει ως αποτέλεσμα να εξουδετερωθεί οποιαδήποτε η εξέλιξη. Θα πρέπει λοιπόν να αυξάνεται και η διάρκεια ζωής του προϊόντος μέσα στη συσκευασία και αυτό φυσικά θα οδηγήσει σε λιγότερη σπατάλη. Και η βιώσιμη λοιπόν εξέλιξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν όλα τα βήματα ληφθούν υπόψη, όλα τα βήματα στην κατανάλωση και στην παραγωγή ενός προϊόντος. Και θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε βήματα προς μια πραγματικά κυκλική οικονομία. τα σκουπίδια ε, στους δρόμους ε, είναι αποτέλεσμα μιας μη συμβατής συμπεριφορά και είναι ε, πραγματικά κάτι πολύ επιζήμιο για το περιβάλλον και επιζήμιο για την ανακύκλωση. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σαφές και κατανοητό προς το καταναλωτή τι είναι το σωστό και πώς πρέπει να συμπεριφερθεί σε ό,τι αφορά τα σκουπίδια του. Τέλος προτείνουμε τα εξή ε, βήματα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές. Καταρχάς, να συνεχιστούν ε, οι εξελίξει των συσκευασιών και θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικότητα των υλικών. Κατά δεύτερον, όπου η ανακύκλωση και η μείωση των υλικών δεν συνάδουν, καλύτερα να υπάρχει μια επιστημονική προσέγγιση του περιφερειακού αντικτύπου, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να λαμβάνουμε ευθύς αποφάσεις που να έχουν ε, νόημα για το περιβάλλον. Κατά τρίτον, να ερευνήσουμε νέε δυνατότητε σε ό,τι αφορά την ε, νέου χρήση και την ανακύκλωση, γιατί είναι πιθανόν, πιθανότατο να υπάρξουν ε, πολλέ εξελίξει και μεγάλη πρόοδο σε ό,τι αφορά την μηχανή ανακύκλωση, όπω είπαν και οι προηγούμενοι μελετέ. Κατά τέταρτον, συνειδητοποιήσουμε τον ε, καταναλωτή και τους εμπλεκόμενους φορές γιατί η έλλειψη κατανόησης ήδη προκαλεί σύγχυση στον καταναλωτή στο μέλλον. Όλες οι δράσεις θα πρέπει τελικά να οδηγούν σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. άλλο ε, ενδεχομένω ο καταναλωτής να μην δεχτεί τα νέα αυτά προϊόντα και αυτό με τη σειρά του θα κάνει ακόμα πιο δύσκολο να πετύχουν τους κοινούς τους στόχους οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική διαπίστωση σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον είναι ότι ο καταναλωτής θέλει και επιθυμεί να κάνει επιλογές πιο φιλικές προς το περιβάλλον στην καθημερινή του ζωή. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για πιο βιώσιμες συσκευασίε. Αυτό δεν θα πρέπει να διακυβευτεί από μια μερική βελτιστοποίηση σε ένα κομμάτι μόνο της αλυσίδας. Θα πρέπει να δούμε όλη τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Τέλος, θέλω να καλέσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους προμηθευτές, τους επιστήμονες, τους πολιτικούς, να μας βοηθήσουν να, καταρτήσουμε, να σχεδιάσουμε καλύτερες συσκευασίε και για το τρόφιμα και για τον καταναλωτή και για το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι κυρίες και κύριοι για την σημαντική αυτή ευκαιρία που μας δώσετε να μοιραστούμε μαζί σας τις απόψεις μας. Ευχαριστώ πολύ, Λεκή Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κύριο Σανταούσκας να λάβει το λόγο για τη δική του παρουσίαση. Καλό σας απόγευμα, ευχαριστώ για αυτή την πρωτοβουλία και για την πρόσκληση. Είναι σκόπιμη και έγκαιρη και όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι έχουμε φτάσει σε μία ε, ισορροπία. Και αυτό γιατί κατά την Παρασκευή για την στρατηγική κάναμε μία ευρύτατη διαβούλευση. Αυτό δεν είναι το πρώτο στρατηγικό έγγραφο για τις πλαστικές ύλες. Ήδη το 2013 υπήρχε το πρώτο πακέτο για τα πλαστικά απορρίμματα που μας έδωσε πολλά στοιχεία από το κοινό και αποτέλεσε ε, πηγή σοφίας για εμάς και μέσα στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας προσπαθήσαμε να ευθυγραμμίσουμε διαφορετικά και συγκρουόμενα πολλές φορές συμφέροντα για να φτάσουμε σε ένα όραμα για το μέλλον. Δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η στρατηγική να ε, εφαρμόσουμε αυτές τις νομοθετικές αλλαγές με την εργαλειοθήκη που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά επιθυμούμε να το κάνουμε. Χτίσαμε αυτή τη στρατηγική σε τέσσερις άξονες ε, η οικονομικός άξονας και πολλά προελέχθησαν για τον τρόπο διαχείρισης των πλαστικών υλών που δεν είναι ευθύς τρόπος διαχείρισης γιατί ήταν ένα βασικό υλικό για την καθημερινή μας ζωή για αρκετές ε, δεκαετίες και έχει αυξηθεί επί 20 φορές τις τελευταίες δεκαετίες. Όμως πρέπει να ελέγξουμε την κατάσταση μετά τη χρήση και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε με ε, ευφύ τρόπο. Δηλαδή όχι μόνο στην παραγωγή του πλαστικού, αλλά τι θα γίνει με το δευτερογενές πλαστικό και πώς μπορεί να επανακάμψει στην πραγματική ζωή. Δεύτερος άξονας, η μόλυνση. Όπως βλέπουμε στις θάλασσες με τα απορρίμματα και παντού. Η κατάσταση δεν είναι υποέλεγχο και ελπίζω ότι οι νόμοι μας και ιδιαίτερα η οδηγία θα κάνουν τη διαφορά γιατί θα θέσουν υψηλότερους στόχους και θα πρέπει να υπολογιστεί σωστά η ανάγκη μας, οι ανάγκες μας ως προς την παραγωγή αλλά και την απόρριψη των υλών. Και θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό έτσι ώστε να μειωθεί η κατάσταση ως προς τα απορρίμματα. Ε, ως προς την καινοτομία θα πρέπει να το δούμε υπό νέα οπτική γωνία, τα πλαστικά, τις πλαστικές ύλες, ε, από τι αποτελούνται, πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτό τον κύκλο έτσι ώστε τα πλαστικά να μην οδηγήσουν σε ε, παράτερη απομάκρυνση. Και επίσης το γεγονός ότι δεν ζούμε μόνοι σε αυτό το πλανήτη, υπάρχουν ε, και άλλες περιφέρειες και όπως βλέπετε η αύξηση γίνεται εκθετικά σε όλες τις περιφέρειες και ό,τι και να κάνουμε ε, δεν ε, είναι αρκετό. Θα πρέπει να ε, δείξουμε ότι έχουμε τις λύσεις και υπάρχουν και άλλες πλευρές, άλλες περιφέρειες του κόσμου που προβάλλουν λύσεις. Αλλά έχουμε μία πλήρη στρατηγική. Θα δράσουμε και με τους τέσσερις άξονες, γι' αυτό θέλουμε τη συμμετοχή της κοινωνίας, των εμπλεκομένων φορέων και γι' αυτό καλωσορίζουμε τις εθελούσιες δεσμεύσεις και τη δράση πολλών ε, βιομηχανιών γιατί έχουμε εκδώσει αυτή την, ε, αυτό το ε, σύγγραμμα για την στρατηγική για τις πλαστικές ύλες για να δούμε τι κάνουν οι βιομηχανίες, τι μπορούν να κάνουν και πώς μπορούμε να δράσουμε για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες να ακολουθήσουν το δρόμο της υψηλότερης βιωσιμότητας. Ε, θα αλλάξουμε δραστικά τον κόσμο, αλλά πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε. Τώρα οι συνάδελφοι έχουν το λόγο. Ο κύριος Φλόρενς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μου έχει προκαλέσει πραγματικά θετική έκπληξη η στρατηγική που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μου αρέσουν αυτά που προτείνει. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς τον τελευταίο εκπρόσωπο της ε, Επιτροπής. Ε, ο Γερμανός Επιτροπός είπε ότι θα εισαγάγει ένα φόρο για τα πλαστικά. Πείτε μας δύο λόγια. Δεύτερο. Έχουμε τώρα την απαγόρευση των κινέζικων εισαγωγών. Αυτό πώς επιτρά. Πού πάνε αυτά τα προϊόντα πάνε σε χωματερές οι οποίες έχουν κλείσει εδώ και καιρό παράνομα. Μία ερώτηση επίσης να κάνω στους συμπεριογνώμονες. Μας είπατε, και αυτό είναι θετικό, ότι υπάρχει η εκ νέου χρήση. Η αξία του προϊόντος διατηρείται ή μειώνεται κατά την ανακύκλωση για την εκπρόσωπο της ΕΦΙΚ, η οποία ευτυχώς και μίλησε τη γλώσσα της, τη μητρική της γλώσσας. Πολύ θετικό αυτό. Για τις ε, δευτερογενείς αγορές. Μήπως όμως στη τελική ανάλυση δεν χρειάζονται πρότυπα όταν γίνεται ανακύκλωση. Εσείς κάνετε ανακύκλωση όσο καλύτερα γίνεται. Αλλά μήπως ε, Αυτό που τελικά χρειάζεται να κάνει ένα κύκλο για να φτιάξει παράθυρα δεν θα αγοράσει τα δικά σας προϊόντα στην περίπτωση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο ε, κύριε Ντάλη λέει η πρόεδρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εσάς που είστε εδώ και αφού συζητάμε το θέμα αυτό. Γιατί προφανώς και απασχολείται ιδιαίτερα το έργο της Επιτροπής μας, γιατί μεγάλε ποσότητε ε, πλαστικού τελικά καταλήγουν ε, στο περιβάλλον και στα ύδατα και στα εδάφη, δημιουργώντας μεγάλο οικονομικό ε, μεγάλη οικονομική και περιβαλλοντική ζημιά και να επικεντρωθώ στο θέμα των σκουπιδιών λοιπόν μιας και πρόσφατα είδα και διάφορες μελέτες του Περιβαλλοντικού Κέντρου στη Γερμανία που αναφέρει ότι 70% της μόλυνσης ε, πλαστικού στους ωκεανούς προέρχεται από 10 ποταμούς και μιλάμε για δεκάδες ε, για πάρα πολλούς ε, τόνους που καταλήγουν στον ωκεανό. Ένα φορτηγό ουσιαστικά κάθε δευτερόλεπτο έχει υπολογιστεί ότι ξεβράζεται στην ε, θάλασσα. Εγώ είμαι από τη Μάλτα και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ένα μεγάλος, μια μεγάλη πηγή μόλυνσης ε, είναι και ο Νείλος. Και σε πολλές περιπτώσεις ε, δυστυχώς η Μεσόγειος θεωρείται μία από τις πιο Μολυσμένε θάλασσε του κόσμου σε ό,τι αφορά τα πλαστικά. Και έτσι λοιπόν θέλω να περάσω στο θέμα των μικροπλαστικών που είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για τη θαλάσσια ζωή και είναι σχεδόν αδύνατο να καθαριστούν τα μικροπλαστικά. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τι απόψει των ε, ομιλητών μα. ιδιαίτερω ε, τη κυρία Μαφρίσλαντ, η οποία σε ό,τι αφορά τα μικροπλαστικά και τις ε, ενδεχόμενες λύσεις καθαρισμού των μικροπλαστικών από τις θάλασσές μας. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι και εμείς δεν θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες ως Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η ρήπανση είναι συνήθως ο βασικός, ε, η βασική αιτία. Να θέσω μια ερώτηση όμως σε ό,τι αφορά τα βιοπλαστικά, τα βιολογικά αυτά πλαστικά, τα βιολογικά πλαστικά αυτά μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία μιας ε, σωστής μετάβασης για τη μείωση των μικροπλαστικών στους ωκεανούς. Όταν μιλάμε για μικροπλαστικά, για βιολογικά πλαστικά μάλλον, μιλάμε για πλαστικά τα οποία μπορούν να διαλυθούν μέσα στις 24 μήνες και μπορούν να επιλύσουν ενδεχομένω το ζήτημα των μικροπλαστικών εν γέννη. Μιλάμε όμως για τη χρήση πλαστικού, και είναι μια μεγάλη πρόκληση. Είναι φυσικά και πρόκληση, αλλά αποτελεί και μια ευκαιρία. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην διαχείριση απορριμμάτων από πολυκρονικό εξοπλισμό, που μπορεί να αποφέρει μεγάλο οικονομικό κέρδος, αν αντιμετωπιστούν σωστά. Επίσης υπάρχει και η τεχνολογία σχεδιασμού για την διαλογή με σωστό τρόπο προκειμένου να είναι πιο εύκολη στη συνέχεια η ανακύκλωση και τα λοιπά πράσινα κριτήρια για την αποσταρμολογήση διαλογή και ανακύκλωση συσκευών. Θα πρέπει τα ζητήματα αυτά λοιπόν τα κοιτάξουμε, να εξετάσουμε το σύνολο της τραγικής και τα πλαστικά να τα αντιμετωπίσουμε συνολικά ως ένα υλικό το οποίο ναι μεν παρουσιάζει προκλήσεις αλλά παρουσιάζει και μακροπρόθεσμα χωρίς το δίχως άλλο ε, και ευκαιρίες. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, ο κύριος Αφρόντα. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να θίξω ένα ιδιαίτερο θέμα, γιατί υπάρχει μια γενική συμφωνία αν και υπάρχουν πολλές αποχρώσεις, πρέπει να μιλήσουμε για την πρόληψη, την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση, το νέο σχεδιασμό και οι σκιώδεις ασχολούνται με την έκθεση του Κοινοβουλίου. Ε, με την ευκαιρία της παρουσίας σας θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι ή προοπτικές για, ως προς ε, τρεις πτυχές. Η παρουσία στα πλαστικά επικίνδυνων ε, ουσιών φενόλης, ας πούμε, ε, ή παραγόγων του χλωρίου που, αντιμετωπίζουν, που αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνες ουσίες. Γιατί έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς γίνεται μετά η αποδόμηση και η ανακύκλωση των πλαστικών. Δεύτερον, ως προς τα μικροπλαστικά, δεν βλέπω και πολλές ε, προοπτικές γιατί η συνάδελφος Νταλή ε, μίλησε για δυσχέρειες. Θα ήθελα να ρωτήσω τον τομέα της ε, βιομηχανίας πέρα από τις μικροπλαστικές ύλες είναι τα μικροπλαστικά που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής και κατά πόσο υπάρχει δέσμευση της βιομηχανίας για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Και τρίτον, πώς βλέπει η βιομηχανία το θέμα των βιοπλαστικών υλών, εάν υπάρχουν προοπτικές, κατά πόσο υποκαθιστούμε το θέμα με ένα άλλο και επίσης, ε, ε, αν απομακρύνουμε τα, τις πλαστικές ύλες από τα ορυκτά, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το θέμα του τομέα. Η κυρία Ντελαή. Κυρία Ντελαή, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι βλέπουμε ότι υπάρχει συνένεση όσον αφορά τη μη χρησιμοποίηση των πλαστικών και αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης τους. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα που δεν θέσαμε. Είναι το θέμα της υποκατάστατής τους από υλικά πιο ανθεκτικά και που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον. Ένα απλό παράδειγμα. Εδώ και κάποια χρόνια λέμε στους ε, παραγωγούς κυπευτικών να μην χρησιμοποιούν πλαστική συσκευασία και χρησιμοποιούν ε, ένα άλλο υλικό. Αυτό θα πρέπει στο μέλλον να το λάβουμε υπόψη. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλαστικά μπουκαλάκια του νερού που θα μπορούσαν αύριο ε, ενδεχομένω να αντικατασταθούν από γυάλινες συσκευασίες ή από μεγαλύτερες ε, ε, συσκευασίες αν θέλετε, παρά αυτά τα μικρά μπουκαλάκια τα οποία καταναλώνουν μεγάλο ποσοστό πλαστικού. Η αποκατάσταση λοιπόν των πλαστικών υλικών από άλλα υλικά που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον είναι κάτι που το έχετε σκεφτεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μποναφέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήδη τέθηκαν πολλές ερωτήσεις Άρα εγώ θα φίξω ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι είναι σημαντικό και θεωρώ σημαντικό. Βλέπω ότι είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία της Επιτροπής διότι και πιστεύω ότι όντως είναι ένα βήμα προς την ε, σωστή κατεύθυνση. Μιλώ για αυτή τη στρατηγική που μας επιτρέπει κυρίως να χειριστούμε δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα να καταπολεμήσουμε την ε, μόλυνση, τη ρήπανση του θαλασσίου χώρου, χώρου πράγμα το οποίο κατά την άποψή μου ακόμη δεν έχουμε αναλύσει τις επιπτώσεις για τις επόμενες γενιές. Τουλάχιστον διεξοδικά δεν το έχουμε κάνει. Δεύτερον, η στρατηγική αυτή μας επιτρέπει να προχωρήσουμε αργότερα προς μία μεταβασή στην κυκλική οικονομία. Διότι σε αυτή την έκφραση υπάρχει το θέμα της, του, του οικονομικού σκέλους. Αν θέλουμε να έχουμε λοιπόν πιο αηφόρο ανάπτυξη, θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη στρατηγική που μας βοηθάει να προχωρήσουμε και να είμαστε καινοτόμοι στα παραγωγικά πρότυπα τα οποία θα ακολουθήσουμε. Βεβαίως, πάντα θα πρέπει να προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε στις προκλήσεις, αλλά να κάνουμε και πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το οποίο θα ήθελα να θέσω στους ειδήμονους είναι το θέμα των πρώτων υλών και των ε, επεξεργασμένων υλών. Πάντα θεωρούμε ότι στην κυκλική οικονομία τα πλαστικά υλικά ή αυτά που θα ανακυκλώσουμε ή όχι είναι σημαντικά. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι ήδη στο πακέτο για την ε, κυκλική οικονομία προβλέψαμε πάρα πολλά μέτρα ε, προληπτικά. Προληπτικά για να αποδείξουμε πόσο έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις για τα θέματα της κυκλικής οικονομίας. Δεύτερον, ο ανακυκλώσιμος χαρακτήρας κάποιων προϊόντων. Πήραμε μέτρα και έχουμε αυξήσει τα ανώτατα όρια ανακύκλωσης και κυρίως σε θέματα πλαστικών. Το πλαστικό έχει γενικά συστατικά, αν θέλετε, σε απόλυτους βαθμούς, τα οποία είναι τα λιγότερο ανακυκλώσιμα σε σχέση με άλλα. Όταν τελειώσει όμως η φάση της ανακύκλωσης, το ανακυκλωμένο προϊόν θα πρέπει να είναι και πιο αηφόρο. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν είναι το εξής. Το αρχικό πλαστικό, η αρχική πλαστική ύλη κοστίζει λιγότερο από την ανακυκλωμένη πλαστική ύλη. Με ποιους μηχανισμούς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία δευτερογενή αγορά πρώτης ύλης από πλαστικό που να έχει μία κάποια αξία στην αγορά. Βεβαίως η διαλογή είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά θα ήθελα να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα αποφασιστικά ε, προς την κυκλική οικονομία. Αν ανακυκλώνουμε προϊόντα τα οποία μετά δεν ξαναχρησιμοποιούμε, δεν πετυχαίνουμε και πολλά πράγματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πεντίτσου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Θα ήθελα παρόλα αυτά να πω κάτι για αυτούς που μίλησαν για τη χρησιμοποίηση και επαναχρησιμοποίηση κάποιων πλαστικών που είναι πάρα πολύ βλαπ βερά για το περιβάλλον ή να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε κάποιες επικίνδυνες ουσίες όπως το βισφενόλ, τα φθαλάτες, πράγματα που είναι θέματα που τα έχουμε συζητήσει ήδη στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρόκειται για επικίνδυνες ουσίες λοιπόν. Στα πλαίσια της έγκρισης του πακέτου για τα απορρίμματα επίσης μιλήσαμε για τη θαλάσσια ρήπανση. Αλλά βεβαίως αυτό δεν επαρκεί, θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Μιλήσαμε για τα μικροπλαστικά, μιλήσαμε για την απαραίτητη έρευνα που πρέπει να γίνει στον τομέα και για τι ενημερωτικέ φύσεις εκστρατεία που πρέπει να κάνουμε για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Ολοκληρώνοντα θα ήθελα να πω το εξή. Πιστεύω ότι η καύση των πλαστικών υλών δεν είναι λύση. Σήμερα Γίνεται λόγος για την παραγωγή θερμότητας από το πλαστικό. Είπαμε ότι μπορούσαμε να υποκαταστήσουμε έτσι διάφορα παραδοσιακά καύσιμα. Η... Τα... Με συγχωρείτε, η καύση όμως είναι κάτι το οποίο εκλείει πολλές, πολύ τοξικές ουσίες στο περιβάλλον. Άρα δεν είναι μία σωστή λύση. Θα ήθελα να μου πει η Επιτροπή ποια είναι η γνώμη της επί του θέματος. Η κυρία Γκροστέτ, κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ανακύκλωση. Μας είπανε ότι 800.000 πολίτες υπέγραψαν υπέρ της ανακύκλωσης, αλλά στα 500 εκατομμύρια τι σημαίνει αυτό. Εγώ στη χώρα μου θα πω το εξής έχουμε προβλέψει διάφορες δυνατότητες διαλογής, ανακύκλωσης, αλλά εδώ και 20 χρόνια δεν έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Πριν από μερικές μέρες έγινε το έξι. Εγώ αγοράζω γάλα σε πλαστική συσκευασία. Αλλάζω παραγωγό και αποφασίζω να αγοράζω γάλα το οποίο ε, παράγουν οι, οι καλλιεργητές, οι γεωργοί στη γειτονιά μου. Και τι μαθαίνω από τον τύπο. Ότι υπάρχει πρόβλημα, διότι το πλαστικό που χρησιμοποιούν για τα ε, μπουκάλες στο γάλα δεν είναι ανακυκλώσιμα. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν αυτό το πλαστικό ήταν πιο φτηνό υλικό. Ε, άρα ξανά παίρνω γάλα μιας μεγάλης βιομηχανικής μονάδας γιατί πρόκειται για πλαστικό ανακυκλώσιμο. Εάν αναφέρω το παράδειγμα αυτό είναι για να δείξω ότι αν υπάρχουν πλαστικά μη ανακυκλώσιμα θα πρέπει να τα απαγορεύσουμε ή να υποχρεώσουμε την βιομηχανία να βρει λύσει. Δεν μπορούμε όμω να συνεχίσουμε να παράγουμε ε, πλαστικό υλικό στη συγκεκριμένη περίπτωση που δεν ανακυκλώνουν. Τώρα υπάρχει η αρχή του όποιος ρηπαίνει πληρώνει. Είναι καταστροφική η θαλάσσια ρήπανση και μας ε, καταπλή... είναι κάτι το οποίο μας αφήνει καταπλήκτους. Πρέπει να βάλουμε τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να παρθούν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, διότι μας δείχνουν Στην Ασία, στον Ειρηνικό, διάφορες τρομερές παραλίες, ονειρικές, αλλά δεν μας δείχνει κανείς το βυθό που βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτές τις παραλίες με τρομερή ρήπανση από τα πλαστικά που συσσωρεύονται. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι δεν έχουμε αρχίσει σωστά την ε, εξέταση και μελέτη του άλλου προβλήματος. Τώρα, ο σχετικός φόρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε τη στρατηγική της τον Ιανουάριο για τις ε, πλαστικές ύλες, αλλά ο κύριος υπεύθυνος υπεύθυνο ε, ε Επίτροπος ε, σε θέματα προπολογισμού μας προτείνει έναν φόρο για να αντισταθμίσει κάτι για το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχουν αμφιβολίες για την εφαρμογή αυτού του φόρου στην Ευρώπη. Θα ήθελα εξαιτήσεις. Λέει ότι θα κάνει επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες πιο ευφυής και πιο ανακυκλώσιμες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει επίσης αυτό που λέγεται για το διαβατήριο του προϊόντος όπου να αναφέρονται τα κύρια χαρακτηριστικά. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματιστικό, είναι κάτι το οποίο είναι αξιόπιστο. Πολλά ερωτηματικά λοιπόν έχω, αλλά πρέπει να πω ότι πραγματικά είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι γιατί στο θέμα αυτό δεν προχωρούμε, περνάει ο καιρός και στο μεταξύ διάστημα αυξάνεται η ρήπανση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε και ο Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς ε, όλους τους συμπεριγνώμονες και προσκεκλημένους μας ε, για τις παρεμβάσεις, γιατί προφανώς ε, σημειώνουμε και όλα αυτά που μας είπατε για την έκθεση θα χρειαστούμε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το είπα. Η στρατηγική αυτή, όπως και περισσότεροι εδώ, θεωρούμε ότι αποτελεί ένα βήμα τεράστιο προς τα εμπρός δεν είναι πλαστικ, ε, στρατηγικά των πλαστικών, δεν επιτρέπεται να είναι κάτι τέτοιο. Μιλάμε για έναν πιο βιώσιμο, και κυκλικό τρόπο αντιμετώπισης ενός πολύτιμου υλικού. Και νομίζω ότι από την άποψη αυτή θα πρέπει να κοιτάξουμε όχι μόνο το ίδιο το υλικό, αλλά Έχουμε υπόψη μας και ενδεχόμενη μετάβαση σε νέα μοντέλα, μοντέλα καταναλωτή, μοντέλα παραγωγής, και e e, κυκλικά για όλο το φάσμα της αλυσίδας παραγωγής και επίσης θα πρέπει να υπάρχει και σύνδεσμος μεταξύ της πολιτικής για τα απορρίμματα, της πολιτικής για τα προϊόντα και της πολιτικής για τα χημικά. Και θα ήθελα να μας πούν οι διάφοροι φορείς και κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς πιστεύουν ότι συγκεκριμένα μπορεί να διαμορφωθεί αυτή η προοπτική. Κατά δεύτερον, συχνά ακούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η νοοτροπία του καταναλωτή, ότι θα πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα. Μπορεί να μην είναι εύκολο, αλλά να ρωτιέμαι. Όταν καθημερινά βλέπω τις διαφημίσεις, το marketing, μα αυτό ακριβώς δεν κάνουν οι παραγωγοί. Επηρεάζουν την συμπεριφορά του καταναλωτή. Και καταφέρνουν λοιπόν να μας πείσουν εμάς ως καταναλωτές ότι ένα προϊόν το οποίο δεν υπήρχε ως τώρα και το οποίο δεν μας έλειπε, ξαφνικά αποτελεί ανάγκη μας. Καταφέρνουν λοιπόν να δημιουργήσουν ε, ανάγκες στον καταναλωτή, μα αν καταφέρνουν τόσο αποτελεσματικά να δημιουργήσουν μια καινούργια ανάγκη, πόσο μάλλον αν ε, ο καταναλωτής προχωρούσε και ε, μπορούσε να, να περάσει στην ένταξη της κυκλικότητας στην μάρκα ενός προϊόντου. Μία ερώτηση για την κυρία Βαράτ, γιατί είπατε ότι οι επικίνδυνες ουσίες αποτελούν ένα πρόβλημα, μια μεγάλη ανησυχία. Είπατε ότι δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε και αναφερθήκατε στη χημική ανακύκλωση. Ισχυρίζεστε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει και στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος αυτού. Και τέλος για την καινοτομία. Νομίζω ότι η καινοτομία πραγματικά θα πρέπει να προωθηθεί, να δοθούν κίνητρα. Σε ποιου τομεί λοιπόν θα θέλατε στην παρούσα φάση να γίνουν κατά προτεραιότητα. Κατά προτεραιότητα επενδύσει σε ό,τι αφορά την καινοτομία προκειμένου για να πετύχει όλη η στρατηγική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά που μας παρουσίασε. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις να κάνω σε ό,τι αφορά και την οδηγία. Για τις ε, ελαφριές σακούλες πλαστικού. Το 2005 λάβαμε, λάβαμε μια οδηγία. Θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον ε, εξετάζεται το ενδεχόμενο απαγόρευση του οξυπλαστικού. Πρόκειται για μία έκθεση και διάφορες μελέτες αναδεικνύουν ότι είναι ακόμα πιο επιζήμιες αυτές οι ουσίες. Μόλι το περιβάλλον δεν μπορούν να συλλεχθούν ε, και αποτελούν μικροπλαστικό. Στην Γεωργία, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ε, χωραφιών και καλλιεργιών φράουλα. Αυτό το ξεπλαστικό, λοιπόν, χρησιμοποιείται και μετά χάνεται πολύ απλά. Χάνεται, αλλά δεν εξαφανίζεται. Είναι καταστροφικό και θα πρέπει να απαγορευτεί. Βιολογικά βιοδιασπόμενα υλικά. Γιατί όλες αυτές οι χρήσεις είναι μονόδρομος. Μπορούμε πολλά να πετύχουμε. Για παράδειγμα, σε διαφορά την ε, οικονομική επιβάρυνση των ε, προϊόντων αυτών σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα πλαστικά μπουκάλια τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Είναι υπηρετά. Δεν μπορούμε λοιπόν να προωθούμε και να αφήνουμε προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να συλλεχθούν στη τελική ανάλυση, να καταλήγουν στα νερά και στα χωράφια μας. Ε, θα πρέπει να είναι πολύ περιορισμένη και απαγορευμένη η χρήση τέτοιων προϊόντων. Αλλά και ο βιομηχανικό κλάδο μα λέει ότι πάντα είναι θετικά διακείμενο, χρειάζονται όμω πιο αυστηρέ προδιαγραφέ για τι πλαστικέ σακούλε. Θα πρέπει να υπολογίσουμε πόσο χρησιμοποιούνται. Γιατί σε ορισμένε περιπτώσει ε, έχουμε την εντύπωση ότι οι κυβερνήσει ε, και η κυβέρνηση στην Δανία θα ήθελα να καταργήσουν και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. αλλά λάβαμε τη μέθοδο υπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά ε, θα πρέπει να λάβουμε τα σχετικά στοιχεία για να σταματήσει αυτή η νοοτροπία ότι εντάξει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το πλαστικό όπως επικρατεί στην ε, Δανία. Θα ήθελα λοιπόν να επικριωθούμε στα πλαστικά μιας χρήσης και να τα αποφύγουμε στο βαθμό του δυνατού. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είμαι εδώ για την παρουσίαση, αλλά θα ήθελα να συνεισφέρω σε αυτή τη συζήτηση για τις πλαστικές ύλες. Κατά την πτήση μου στις Βρυξέλλες ε, χρησιμοποίησα πλαστικά μίας χρήσης. Το φλιτζάνι μου, τα μαχαιροπύρουνα, τα, το δίσκο, και ούτω καθεξής. Και τα πλαστικά μπουκάλια βεβαίως. Άρα και εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Θέλουμε να μειώσουμε τη χρήση πλαστικών, αλλά πολλές φορές το χρησιμοποιούμε για τη διατήρηση για τη συντήρηση των τροφίμων. Άρα πολλές πολιτικές είναι αμφίσιμες και συγκρουσιακές. Προσπαθώ να ανακυκλώνω πάντα, αλλά με τα πλαστικά χάνω το παιχνίδι γιατί προσπαθώ να πλένω τα πλαστικά για να μην περιέχουν ύλες που είναι μολυσματικές, αλλά καταναλώνω νερό για να το κάνω αυτό. Ένας τομέας που χρησιμοποιεί τις πλαστικές ύλες είναι ο τομέας της ε, γεωργίας και ο ποροκυπευτικών. Αλλά θα πρέπει να δούμε πού πάνε αυτά τα πλαστικά και θα πρέπει να βρούμε ένα υποκατάστατο. Άρα για την βιοοικονομία που είναι μέρος της κυκλικής οικονομίας, ε, η βιοοικονομία είναι η λύση ίσως του προβλήματος. Πολλοί είσαστε αποκαρδιωμένοι. Αλλά το ότι λάβαμε απόφαση ως προς την Κίνα σημαίνει ότι συνειδητοποιούμε το πρόβλημα, ενώ στη χώρα μου, στην Ιρλανδία, δυστυχώς είμαστε οι μεγαλύτεροι χρήστες πλαστικών, άρα υπάρχει μια συνειδητοποίηση του προβλήματος, κάτι το οποίο κάνει πολύ καλό. Τελειώνουμε με τον κατάλογο ομιλητών και θα ήθελα η Επιτροπή και οι εμπλεκόμενοι φορείς να λάβουν το λόγο και να συνεισφέρουν στη συζήτηση όπως εξελίχθηκε. Θα ακολουθήσουμε την ίδια σειρά. Την ίδια σειρά, λοιπόν. Η κυρία Βάλρετ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και έχω πολλές ερωτήσεις να απαντήσω. Ακούσαμε διάφορε ερωτήσει για τα βιοπλαστικά, τα βιολογικά πλαστικά. Κατά πόσο αποτελούν τη λύση, κατά πόσο μπορούν να συμβάλλουν πραγματικά για καλύτερη αντιμετώπιση των ε, πλαστικών. Θα πρέπει να γίνει μια διάκριση. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των βιοδιασπόμενων και των βιολογικών πλαστικών, δηλαδή πλαστικών που προέρχονται από βιολογική προέλευση. Και τα υλικά τα οποία προέρχονται από βιολογικές ε, πηγές δεν είναι απαραίτητα βιοδιασπόμενα. Γιατί, γιατί βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται για παράδειγμα βιομάζα για να δημιουργηθούν αντίστοιχα προϊόντα, αντίστοιχα με πλαστικά από την πετροχημική βιομηχανία. Αυτά όμως δεν είναι βιοδιασπόμενα, άρα δεν θεωρώ ότι αυτή η λύση απαραίτητα είναι ιδανική. Υπάρχουν διαδιασπόμενα υλικά αλλά δεν μπορούμε να τα εξισώσουμε όλα μεταξύ του. Υπάρχουν δύο πλαστικά τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν προκειμένου να είναι βιοδιασπόμενα. Αυτά έχουν την αξία του, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε πώ τα αντιμετωπίζουμε. Και αυτά θα πρέπει να συλλέγονται διαφορετικά. Γιατί αν αυτά τα βάλουμε μαζί με τα υπόλοιπα πλαστικά και ακούσαμε πόσο δύσκολο είναι να γίνει η διαλογή των υλικών για την ανακύκλωση. Αν λοιπόν τα βιοδιασπόμενα καταλήξουν με τα άλλα πλαστικά, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Μας δημιουργείται πιο πολλά προβλήματα και τελικά είναι λιγότερο αποτελεσματική ανακύκλωση. Και έτσι μειώνεται η ποιότητα. Δεν είναι λοιπόν προφανής η λύση, αλλά προφανώς θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε τις επιλογές που κάνουμε. Άκουσα και πολλές ερωτήσεις για την παρουσία ανησυχητικών ουσιών και τις ανησυχίες που επικρατούν. Όντως, στην παρουσίασή μου λοιπόν είπα ότι η ύπαρξη ανησυχητικών ουσιών μπορεί να επιληθεί ενδεχομένως μέσω χημικής ανακύκλωσης. Υπάρχουν δυνατότητες για να επιληθούν τέτοια ζητήματα και να αφαιρεθούν οι επιζήμιες και ανησυχητικές ουσίες. Και για την εκ νέου χρήση των αρχικών πολυμερών υπάρχουν διάφορες ανησυχίες για τα θερμοσέντ ό,τι αφορά τη χημική τους ανακύκλωση και κάποιοι λένε για τα μονομερή τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη χρήση άλλων χημικών. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση και για το μέλλον για την αφαίρεση των SWHS. Αλλά σίγουρα θα σημαίνει αυτό παρετέρω επενδύσει σε καινοτομικά προϊόντα. Έχουμε κάνει μεγάλο δρόμο, έχουμε διανύσει σε επίπεδο εργαστηρίων, έρευνα. Τώρα πρέπει να περάσουμε βέβαια στο επίπεδο τη επένδυση και της επένδυσης σε μεγάλες ε, εγκαταστάσεις. Αυτό λοιπόν σίγουρα αποτελεί μια πρόταση. Αν ζητάτε επενδύσεις στην καινοτομία, θεωρώ ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα της χημικής ανακύκλωσης. Θα είναι κρίσιμο. Τέλος, να επανέλθω στο SVHS, ε, το υλικό αυτό και η ύπαρξη τέτοιων ανησυχητικών ε, ουσιών δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δεν μπορούν να κυκλοθούν. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μια προσέγγιση βάση αξιολόγηση κινδύνου. Να μην κοιτάμε τόσο πολύ του κινδύνου, αλλά τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται ο άνθρωπο Και διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τα ανακοινοκυκλωμένα αυτά α, υλικά χρησιμοποιούνται εκ νέου και αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει ε, Κίνδυνο και ότι τα ωφέλη είναι πιο πολλά από ότι τα μειονεκτήματα, θεωρώ ότι μπορούν να κυκλοφορούν και τα προϊόντα αυτά. Και η οδηγία REACH για παράδειγμα, η οποία είναι σαφέστατη. Θεωρούμε ότι θα γίνει μια σωστή ε, αξιολόγηση και στην ε, επιστημονική αλλά και στην κοινωνικο-οικονομική επιτροπή για να δούμε κατά πόσο να αξίζει τον κόπο και κατά πόσον μπορεί να γίνει ανακύκλωση. Και πρέπει να γίνει ανακύκλωση και βλέπουμε ότι έχουν δοθεί πάρα πολλέ ε, άδειε προ την κατεύθυνση αυτή σήμερα και ότι αν ακολουθήσουμε την ίδια επιστημονική προσέγγιση, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για άλλα πολλά υλικά. Ευχαριστώ. Για να δω έγινε και μία ερώτηση για ενδεχόμενα διαβατήρια υλικών, κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό και εφαρμόσιμο και σκόπιμο. Κοιτάξτε, υπάρχει μία ανησυχία μεταξύ των υπεύθυνων ανακύκλωση για το κατά πόσο ανακυκλώνονται κάποια υλικά και φυσικά χρειάζονται σωστή επικοινωνία σε όλη την αλυσίδα παραγωγής μέχρι σε το σημείο που τελικά το υλικό καταλήγει στον καταναλωτή, όπου χάνονται πολλές πληροφορίες, γιατί τελικά το προϊόν αυτό καταλήγει πάλι στα σκουπίδια. Και τελικά θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσον υπάρχουν ανησυχητικές ουσίες στα προϊόντα. Δεν είμαστε πεπισμένοι ως κλάδος ότι χρειάζεται μια τέτοια διαβατήρια για τα υλικά. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές σύγχρονες ε, τεχνολογίες όπως η blockchain η οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ενδεχόμενη λύση. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνουν επενδύσει για να δούμε το πώς ε, μπορούμε να πετύχουμε καλύτερη επικοινωνία σε όλη την γάμα της αλυσίδας παραγωγής. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα τα αφήσω στους συναδέλφους να τα απαντήσουν. Ευχαριστώ, Λέκη Πρόεδρος. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα ήθελα να δω το θέμα των μικροπλαστικών. Δεν υπάρχει περίπτωση καθαρισμού όταν βρίσκονται στους ωκεανούς θα βυθιστούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν επιπτώσεις, γιατί θα αλλάξει η ποιότητα του βυθού σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε τα μικροπλαστικά από το να μπαίνουν στους ωκεανούς. Τώρα, ως προς τα βιοπλαστικά και τα πλαστικά που μπορούν να αποδομηθούν. Δεν υπάρχουν ε, διεθνείς συμφωνίες, είναι νέα υλικά και αυτό που έχει σημασία είναι η αποδόμηση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Δηλαδή στο, στα ποτάμια και στη γη δεν υπάρχει αποδόμηση. Μιλάμε για ένα 10% υλικού το οποίο δεν αποδομείται. Επειδή λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, είμαστε και πολύ ανήσυχοι ως προς την πίεση υπέρ των βιοπλαστικών. Έχουν ε, ε θετικές επιπτώσεις, αν και θα πρέπει να ξέρουμε πώς να συλλέγουμε αυτά τα υλικά στο τέλος της ζωής τους. Πώς ορίζουμε τη βιωσιμότητα. Μιλήσαμε για βιώσιμα υλικά και η βιωσιμότητα είναι κάτι το πολύ διαφορετικό για τον καθένα. Όταν μιλάμε για βιωσιμότητα, δεν θα πρέπει να μιλάμε για τα παροδυσιακά συστήματα διαχείρισης λιμάτων. Αυτό ισχύει και όταν μιλάμε για διάφορες μορφές επεξεργασίας, γιατί ορισμένες μορφές ανακύκλωσης δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον όταν μιλάμε για κατανάλωση ενέργειας και η ανακύκλωση δεν είναι η απάντηση για όλα, δεν είναι πανάκια, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πυρόληση, χημικές ουσίες κλπ. Μιλήσαμε για την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών σήμερα. Όπως είπε και ένας ευρωβουλευτής, είχαμε πολλές εκστρατείες ε, συμπεριφοράς, αλλά είναι καλύτερα να δίνουμε τις εύκολες λύσεις στους πολίτες. Θα πρέπει όλα να γίνουν πιο εύκολα με την επαναχρησιμοποίηση. Εκεί όπου υπάρχει επαναχρησιμοποίηση ε, φιαλών, τότε οι πολίτες επιστρέφουν τις ε, φιάλες αυτές. Γιατί να μην υπάρχουν συστήματα λοιπόν επιστροφής και απόθεσης. Νομίζω ότι υπάρχει δραστική αλλαγή συμπεριφοράς, το βλέπουμε με τις πλαστικές σακούλες και ίσως θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να τρώνε μέσα σε ένα εστιατόριο, όχι να, να χρησιμοποιούν το take away. Θα πρέπει να μειώσουμε την χρήση του πλαστικού. Αυτό είναι ανώτερη ανάγκη για να μειώσουμε βεβαίως και την παρουσία τους στο θαλάσσιο περιβάλλον και στο οικοσύστημα, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ε, όταν έχουν ε, μακρά ζωή και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην, ε, στις ΗΠΑ γίνεται λόγος για 264, 264 μονάδες ε, δημιουργίας πλαστικών υλών. Άρα μπορούμε να έχουμε αύξηση κατά 20% των πλαστικών. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα πλαστικά εκεί που είναι αναγκαία και εκεί που υπάρχουν ευεργετήματα για το κλίμα και το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάγγελούδε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν τόσα πολλά θέματα τα οποία άκουσα και θα ήθελα να αρχίσω με το πόσο σημαντικό είναι να δούμε ποιος είναι ο στόχος της κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή να μειωθούν οι εκπομπές ε, ε, ε, διοξιδίου του άνθρωπος και να διασφαλίσουμε τους πόρους που διαθέτουμε. Ακούω να γίνεται συζήτηση για τα βιοπλαστικά ή για τις εναλλακτικέ λύσεις. Πρόκειται για θέματα που μπλέκονται μεταξύ τους και είναι δύσκολο να βρούμε λύσεις. Επιτρέψτε μου να μιλήσω για κάποια θέματα ε, είπε κάποιος ότι η κυκλικότητα δεν θα σώσει το πρόβλημα. Η κυκλικότητα θα αυξήσει την αποδοτικότητα των πόρων και χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους και θα πρέπει να τις χρησιμοποιούμε πιο έξυπνα. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε χρησιμοποιώντας καλύτερα τα πλαστικά για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές ε, ρήπων διοξυδίου του άνθρωπος. Αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε ε, Βεβαίω ε, λέγεται ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε το πλαστικό με άλλα υλικά. Γιατί μόνο τα πλαστικά. Ε, και πολλά άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται και πιστεύουμε ότι τα χρειαζόμαστε στην κοινωνία μπορούμε να αντικαταστήσουμε. Ας δούμε τις, μια πρόσφατη μελέτη για το πραγματικό κόστος Εάν ε, αντικαταστήσετε σφαιρικά το πλαστικό με άλλα υλικά, θα αυξηθεί το ε, κόστος και το άχθος για το περιβάλλον. Δεν μπορεί λοιπόν ε, να κάνουμε αποσπασματικά τέτοιου είδους αντικαταστάσεις υλικών. Όπως σας είπα για την κυκλικότητα είναι σημαντικά άλλα πράγματα. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι έχουμε τόσο πολύ ενισχύσει τον ε, πυλώνα της ε, πρόληψης και δεν έχουμε ίσως κάνει πάρα πολύ καλή διαφήμιση για την καλή χρησιμοποίηση των πλαστικών. Τώρα, θα πρέπει να αυξήσουμε περισσότερο την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση και την ε, παράταση του κύκλου ζωής κάποιων πλαστικών ειδών. Φερρυπίν. Έχετε με ένα πλαστικό μπουκάλι νερού, το οποίο είναι ανακυκλωμένο και άλλο δεν είναι. Αυτή εδώ ε, είναι ανακυκλωμένο που κρατάει η ομιλήτρια και μας δίνει πολύ καλής ποιότητας νερό υπάρχει και το καπάκι. Θα επανέλθω αργότερα. Το, ε, το μπουκαλάκι γίνεται από πλαστικό το οποίο το λέμε πιτί. Γιατί, διότι είναι ένα εύπλαστο υλικό το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιηθεί. Στην καινοτομία λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα συστήματα διαλογής, επαναχρησιμοποίησης, επανακύκλωσης και καλής επανακύκλωτης επανακύκλωσης ε, είναι κάτι το οποίο γίνεται συστηματικά. Πολύ καλή δουλειά θα πρέπει να γίνει. Άρα αυτό το υλικό που έχω στα χέρια μου είναι πολύ καλής ε, ποιότητας. Και βεβαίω πολλά πλαστικά ανακυκλώνονται, αλλά θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατικό τρόπο και καλύτερα. Γι' αυτό μίλησα εγώ για τον ε, ε, οικολογικό σχεδιασμό. Όλα αυτά ώστε να μπορέσει ε, να υπάρχει κυκλικότητα και αηφόρος χρησιμοποίηση. Κάτι άλλο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Όπως σας είπα, κυκλικότητα, δεύτερον, στο θέμα των απορριμμάτων. Ας μην ε, τα συγχαίουμε τα θέματα αυτά. Λοιπόν, δυστυχώς, στα απορρίμματα πηγαίνουν τα καπάκια. Θα μπορούσε κανείς ότι είναι πολύ μικρό το καπάκι σε σχέση με το μπουκαλάκι. Υπάρχουν όμως καπάκια τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο κολλημένα στη συσκευασία. Και έτσι ε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο καταναλωτής τα πετάει τα καπάκια όπου βρει. Βλέπετε, υπάρχει κάτι το διαφορετικό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει με καινοτόμο βλέμμα να το κοιτάξουμε. Πρόσφατα διάβασα ότι θα πρέπει όλες τις πλαστικές συσκευασίε να τις καταργήσουμε. Γιατί, για ποιο λόγο. Εγώ χρησιμοποιώ σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην ε, κατάψυξη έχουμε ε, προϊόντα ε, κατεψυγμένα τα οποία για καλό λόγο είναι σε πλαστική συσκευασία μίας χρήσης. Πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και όταν τα αποψύξω πετάω το πλαστικό. Θα πρέπει όμως και αυτού του είδους το πλαστικό να μπορέσω να το ανακυκλώσω. Αυτού του είδους τα πλαστικά προ μίας χρήση, δεν είναι μίας χρήση για τα κατεψυγμένα προϊόντα. Μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε. Άρα θα πρέπει να ενημερωθούμε καλύτερα. Θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αυτό το ακούω συχνά, ότι όλα αυτά τα συγχαίουμε λίγο. Τώρα, το, τα βιοπλαστικά, η κυκλικότητα, θα πρέπει να μπορέσουμε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε άλλου είδους πρώτες για να κάνουμε ε, βιοπλαστικά. Ε, ίσως ανανεώσιμες πρότεσίλες. Όλα αυτά για να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των υλών που χρησιμοποιούμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε κατά νου και θα πρέπει με την εξέλιξη της επιστήμης να προχωρήσουμε. Ένα τελευταίο στοιχείο για τα μικροπλαστικά. Όντως, τα μικροπλαστικά όταν δημιουργηθούν στο περιβάλλον δύσκολα θα μπορέσουν να ε, απομακρυνθούν. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ πραγματιστές και προσεκτικοί ώστε να μην δημιουργούνται αυτού του είδους τα μικροπλαστικά και όλα αυτά τα πλαστικά τα οποία ε, απορρίπτονται στην θάλασσα κυρίως. Επίσης, πρέπει να πω ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, καλύτερη ενημέρωση για τα μικροπλαστικά, καλύτερη έρευνα με καλύτερη χρηματοδότηση και έχουμε δει αρκετές μελέτες για το θέμα, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε. Διότι τα πλαστικά δεν είναι μέρος του περιβάλλοντος, δεν πρέπει να βρίσκονται μέσα στο περιβάλλον, άρα πολλές δράσεις είναι δυνατόν να ληφθούν. Το μήνυμά μου, παρακαλώ, βοηθηθείτε ενημερωθείτε. Ένα θέμα αφορά την ε, κυκλικότητα και την ε, ε, παραγωγή προϊόντων χαμηλού επίπεδου εκποδών διοξιδίου του άνθρακος και άλλο θέμα είναι αυτό της αποδοτικής χρησιμοποίησης των υλικών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μακηματήλα, νομίζω ότι απαντήθηκαν οι περισσότερες ερωτήσεις θα ήθελα να σταθώ μόνο σε ορισμένα σημεία. Σε σχέση με τις επενδύσεις πιστεύω ότι δεν υπάρχει η μοναδική καλύτερη λύση για επενδύσεις. Ό,τι φέρνει καλά αποτελέσματα στην όλη διαδικασία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Υπήρχαν ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με τους καταναλωτές και Πράγματι, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβούν στη σωστή επιλογή. Είτε πρόκειται για ανακύκλωση, είτε επαναχρησιμοποίηση, είτε πρόληψη. Ό,τι είναι καλύτερο για το περιβάλλον είναι καλύτερο και για τον καταναλωτή. Τη στιγμή που αυτό γίνει κατανοητό μέσω στοιχείων ως προς τα μικροπλαστικά πιστεύω ότι χρειάζεται έρευνα για να θέσουμε προτεραιότητες αν ε, αναλυφθεί η δράση πριν από την έρευνα, τότε δεν θα γίνει τίποτα έμπρακτα. Ως προς τα απορρίμματα, ναι, θα πρέπει να γίνεται η συλλογή τους, χρειάζεται καλή εκπαίδευση, όπως είπα και ο προηγούμενος, προηγούμενη ομιλήτρια και ως προς την βιωσιμότητα θα πρέπει να έχουμε εναρμονισμένα κριτήρια Διαφορετικά θα, ε, δεν θα υπάρξει η απλούστευση που ορίζει η ανάγκη της βιωσιμότητας. Σας ευχαριστώ όλους. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σαουντάσκας αν έχει κάτι να μας πει από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων Νομίζω ότι θίξαν όλες τις πτυχές οι ευρωβουλευτές καθώς και οι πάνελιστ. Οι εμπλεκόμενοι φορείς μας, ε, ενδιέφερε, μας ενδιαφέρει η στρατηγική στο σύνολό της και φυσικά το θέμα του τέλους είναι ύψης της σημασίας θα μας απασχολήσει μέσα στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής και θα δούμε ποια θα είναι τα ε, φορολογικά μέτρα που ενδείκνυνται. Βεβαίως μας απασχολεί το θέμα. Είναι πολύ ευαίσθητο, αλλά δεν θέλουμε να ανακύψουν ζητήματα τα οποία δεν έχουμε σκεφτεί επαρκώς αλλά φυσικά ε, μας απασχολεί το θέμα, το εξετάζουμε. Σε σχέση με την απαγόρευση προϊόντων από την Κίνα, θα ήθελα να πω ότι και η Κίνα προχωράει με τις απαγορεύσεις, κάτι το οποίο οδηγεί σε μία αναχέτηση του εμπορίου ως προς τα απορρίμματα. Εδώ και χρόνια μου αναφέρει η βιομηχανία διαχείρισης λιμάτων ότι ένα από τα προβλήματα που είχαν ήταν να γνωρίζουν πού πάνε τα απορρίμματα που φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι χάνουμε υλικό προς τρίτες χώρες. Τώρα είναι, έχουμε την ευκαιρία να το πάρουμε πίσω αυτό το υλικό, αλλά θα πρέπει να μην το καταστρέψουμε. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι η αποτέφρωση είναι η δεύτερη χειρότερη λύση στην ιεράρχηση. Δεν θα πρέπει να την ενθαρρύνουμε. Η αποτέφρωση είναι καλή όταν ε, δεν υπάρχει πιθανότητα ανακύκλωσης, αλλά αυτό αποτελεί εξαίρεση. Επίσης ε, θα ήθελα να υποστηρίξω τις ε, δηλώσεις για την τυποποίηση. Η τυποποίηση είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι θεωρούσαμε. Υπάρχει θέμα προδιαγραφών ε, βιοαποδόμησης, γιατί αυτό σημαίνει κάτι διαφορετικό ανάλογα με τις γεωγραφικές παραμέτρους και το κλίμα. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο. Το ίδιο αφορά και τις προδιαγραφές για την συλλογή πλαστικών απορριμμάτων. Γιατί η βιομηχανία θέλει να επαναφέρει αυτά τα πλαστικά στην παραγωγή, αλλά θα πρέπει να έχουμε πολύ καλή πρώτη ύλη από τα δευτερογενή ε, πλαστικά. Θα πρέπει δηλαδή να είναι σίγουρη και ασφαλής η χρήση, η χρήση τους. Ως προς τις χημικές ουσίες θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει και μία νέα ανακοίνωση εξίσου σημαντική για την ε, διάδραση αυτή και τα χημικά προϊόντα ως απορρίμματα. Υπάρχουν πρακτικά ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τους οικονομικούς φορείς, γιατί λένε ότι υπάρχουν χάσματα και επικαλύψεις που θα πρέπει να μας απασχολεί. Και επίσης τι γίνεται με τις ύλες που κληροδοτούμε αλλά ε, τι γίνεται σε αυτή, στην περίπτωση απορριμμάτων που ε, μπαίνουν στον κύκλο, πρέπει να μπουν στον κύκλο ή να βγουν από τον κύκλο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η νομοθεσία μας για τις χημικές ουσίες είναι καινοτόμος είτε πρόκειται για πλαστικά είτε για άλλα υλικά ε, έχουμε καθαρά υλικά που ξαναμπαίνουν στην οικονομία. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τις ε, καλύτερες δυνατές λύσεις ως προς την ε, ε, οξιαποδόμηση. Θεωρώ ότι στο Ελσίνκι μιλήσαμε για τους περιορισμούς και ε, πρόκειται για μια διαδικασία που είναι πιο γρήγορη από την συναπόφαση και πιστεύω ότι ο οργανισμός αυτός θα δράσει με, τη, με τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές. Αυτό αφορά και τα μικροπλαστικά, τα οποία ενσωματώνονται σε προϊόντα και το REACH θα μπορέσει να αποτελέσει μία γρήγορη λύση. Τα βιοπλαστικά μπορούν να δημιουργηθούν και από την κλωστοϊφαντουργία και θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά αυτό το θέμα. Αυτά είναι τα περισσότερα από τα στοιχεία που θα ήθελα να θίξω και σας ευχαριστώ για αυτή την ενθαρρυντική συζήτηση. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Πολύ, σας ευχαριστώ όλους. Βρίσκομαστε στην αρχή αυτής της συζήτησης. Σας καλώ να συνεχίσετε και σε άλλες συνεδριάσεις. Ευχαριστώ πολύ τις, όλους για τη συμμετοχή τους, τους εκπροσώπους των φορέων όλους τους συμμετέχοντες. Σας ευχαριστώ. Λίγη η σημερινή μας συνεδρίαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι την Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι με την Πέτη, την Πέμπτη, πάει μια κοινή ακρόαση. Ευχαριστώ.